Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ο συνάδελφός μας ο κύριος Μακμίλαν Σκοτ θα έπρεπε να ξεκινήσει τη συνεδρίαση τη συνεδρίασή μας αλλά αυτή τη στιγμή είναι εμποτιλιασμένος στις Βρυξέλλες μαζί με τον Πολ Μακκάρτνεϊ. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο Έντουαρτ με τον Πολ αλλά θα πρέπει εμείς να ξεκινήσουμε χωρίς την παρουσία του. Ήταν η δική του πρωτοβουλία να προσκαλέσει τον Σερ Πολ Μακάρνι και επίσης και τον κύριο Πατσάουρη, ο οποίος είναι μαζί μας εδώ, ώστε να ξεκινήσουμε την ακρόαση αυτή για την κλιματική αλλαγή και την τροφιμική ασφάλεια. Ξέρουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα την επόμενη εβδομάδα λαμβάνει η χώρα η διάσκεψη της Κοπενχάγης. Όλος ο κόσμος είναι στην Κοπενχάγη. Είναι πάρα πολύ λοιπόν ε, σημαντική χρονική στιγμή για την συνεδρίασή μας σήμερα. Τι διακυβεύεται στην Κοπενχάγη. Η διαπραγμάτευση <clears throat> παγκοσμίων δεσμευτικών συμφωνιών για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή. Δεν πρέπει να περιορίσουμε τις προσδοκίες μας. Πρέπει να τις πραγματοποιήσουμε τις προσδοκίες μας. Ξέρουμε ότι ο χρόνος κινείται εναντίον μας. Πρέπει να είμαστε λοιπόν Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν την κλιματική αλλαγή και η Ευρώπη έχει παρουσιάσει το πιο φιλόδοξο πακέτο που περιλαμβάνει δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, εμπορία εκπομπών, μείωση των εκπομπών από μέσα μεταφορών, κατανομή προσπαθειών. Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν με χρηματοδότηση κτλ. έχουν υποστηριχθεί από το Κοινοβούλιο και από την Κομισιόν. Όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ σημαντική συμβολή και ένα σαφές μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει σοβαρά τις υποχρεώσεις της. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα για τη διάσκεψη της Κοπεχάγης με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων. Θέλουμε να τονίσουμε ότι συλλογικά οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 25 με 40% μέχρι το 2020, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες να φτάσουν να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 15-30% σε σχέση με το λεγόμενο σενάριο business as usual, δηλαδή το τι θα γινόταν χωρίς κανένα μέτρο. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύει την αλληλεγγύη της με τον αναπτυσσόμενο κόσμο, γιατί η συνολική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή και την μείωση των εκπομπών δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 30 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030. 5 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα πρέπει να είναι η αρχική χρηματοδότηση στις χώρες αυτές και στη συνέχεια θα πρέπει να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα ποσά αυτά. Αυτά είναι θέματα λοιπόν αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αρχίσει να τακτοποιεί τα του οίκου της. Θα χρειαστεί να πετύχουμε τους στόχους του Κιώτο από το 1997 που θεωρούμε ότι θα τους επιτύχουμε με μεγάλη άνεση. Κυρίε και κύριοι, είναι καιρό επιτέλους η διεθνής κοινότητα να επομιστεί τις ευθύνε της και να συνεργαστεί μαζί μας για να μπορέσουμε να ξέρουμε κοινέ λύσει. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Χαιρετίζουμε την προσωπική δέσμευση του κ. Ομπάμα για, και σε εθνικό επίπεδο στις Πολιτείες και για μια επιτυχία στην Κοπενχάγη. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι ήδη η Κίνα έδειξε τη δέσμευσή της προτείνοντας να μειώσει στο τωρινό της πενταετές σχέδιο την ένταση ε, ενέργειας κατά 20%. Και η βασική ομάδα στις, ε, στη Σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή, η Ινδία, η Κίνα και άλλες χώρες, προετοιμάζουν ένα εναλλακτικό κείμενο εναντί αυτού που προετοίμασε η κυβέρνηση της Δανίας. Όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία. Αυτό το κείμενο έχει και την υποστήριξη των ε, 77 χωρών, των G77, που πράγματι επιζητούν μια σοβαρή συζήτηση για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, θέλω να τονίσω και ένα άλλο σημαντικό σημείο. Υπάρχει ανάγκη να έχουμε μια πραγματική ενεργειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πολλούς είναι σημαντικός ο αγώνας για την κλιματική αλλαγή, και φτάνουν τα πράγματα ως εκεί. Αλλά για άλλους τα θέματα της ενέργειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την ενεργειακή ασφάλεια τροφοδοσίας, γιατί τους είναι απαραίτητη. <clears throat> Χωρίς μια πλήρη συνολική πολιτική ενέργειας που να περιλαμβάνει και την ασφάλεια εφοδιασμού δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή κοινότητα ενέργειας. Χρειαζόμαστε μια νέα αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά την παραγωγή, διανομή και κατανάλωση ενέργειας. Χρειαζόμαστε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές για τον 21ο αιώνα στον τομέα της ενέργειας και να εξασφαλίσουμε νέους ενεργειακούς πόρους χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος κτλ. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί από μόνο του να αποφύγει να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Φυσικά κανένα κράτο μέλο δεν έχει του οικονομικού πόρου να αναπτύξει όλε αυτέ τι ενεργειακέ πηγέ μόνο του. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μονάχα με συνεχεί ευρωπαϊκέ επενδύσει σε μακρόπνο επίπεδο. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα περιλαμβάνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, την έννοια τη αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά την παροχή ενέργεια και την ενεργειακή πολιτική. Η αλληλεγγύη αυτή σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια κοινότητα <clears throat> που θα πρέπει να οικοδομήσει ένα χώρο αλληλέγγυο σε σχέση με την ενέργεια και χώρο χαμηλών εκπομπών. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη θα είναι ένα σημαντικό παίκτη στο παγκόσμιο στερέωμα για του στόχου τη κλιματική αλλαγή. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο άνθρωπο θα βρίσκεται σε ειρήνη πια με τον πλανήτη. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε σαν άτομα, ο κάθε ένας από εμά. Εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή απαιτείται και μια αλλαγή στις συνήθειές μας. Από τον τρόπο που οικοδομούμε τα σπίτια μας, από τα αυτοκίνητα που οδηγούμε, από τα εργοστάσια τα οποία κατασκευάζουμε και φτάνοντας μέχρι τα αντικείμενα και τα είδη που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Καλύτερη μόνωση των ε, κτηρίων, καθαρότερα καύσιμα, Όλα αυτά είναι απαραίτητα γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε ρεαλιστικά τους στόχους που θέλουμε να έχουμε. Θα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος ζωής μας. Ο τρόπος με τον οποίο διατρεφόμαστε. Δεν θέλουν όλοι να είναι χορτοφάγοι. Η κόρη μου είναι χορτοφάγα τα τελευταία δέκα χρόνια. Εγώ όχι. Αλλά όλοι μας μπορούμε να σταματήσουμε να τρώμε κρέας για μία μέρα τη βδομάδα. Είναι μια εκκίνηση, μια πολύ καλή ιδέα που έχει προωθήσει ο Πολ Μακάρτνε, ο οποίος σε λίγο θα είναι μαζί μας. Λιγότερο κρέας σημαίνει λιγότερη θερμότητα. Ίσως δεν θα έχουμε κάθε μέρα μια μέρα όπως σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σήμερα πρέπει να πω ότι τα μισά πιάτα στο εστιατόριο των ευρωπαϊκών, στα εστιατόρια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι χωρίς κρέας. Η πρωτοβουλία για μια Δευτέρα χωρίς κρέας είναι μια πρωτοβουλία που επιτρέψει στους πολίτες να επιφέρουν μια ουσιαστική αλλαγή. Να μειώσουμε την υπερπαραγωγή του κρέατος στον κόσμο μας. Πρέπει να δράσουμε συνολικά για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες αυτές αλλαγές. Δεν μπορούμε όμως να παραγνωρίσουμε αυτά τα οποία κάνουμε στο τοπικό επίπεδο, στο σπίτι μας, στον τόπο εργασίας μας, τι προσωπικές μας συνήθειες. Υπάρχει ένα γνωστό τραγούδι των Beatles και αν το παραφράσω λιγάκι, έλεγε «Έρχεται ο ήλιος, here comes the sun». Ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε ότι θα μπορούμε να το επαναλάβουμε αυτό και στο μέλλον. Σιγά σιγά λιώνουν οι πάγοι, θα πρέπει να βγει ο ήλιος μέσα από την αχλή του χειμώνα και να εξασφαλίσουμε ότι it's all right, ότι όλα πάνε καλά. Καλή τύχη στον πλανήτη μας. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. ο ε, Ευρωβουλευτής Μακμίναν Σκοτ. Παρά ο πρόεδρος Μπούσεκ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Έντουαρτ Μακμίναν Σκοτ, που προτείνατε και το Προεδρείο δέχτηκε. Οι συνάδελφοί μου αντιπρόεδροι και εγώ δεχτήκαμε την υπέροχη ιδέα σας να προσκαλέσετε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σερ Πολ Μακάτνεϊ και τον Μισελ Πατσάουρη που είναι ε, ο υπεύθυνο για θέματα κλίματος στα Ενωμένα Έθνη. Όλοι εδώ ε, αναμένουμε την έλευση των προσώπων αυτών. Έχετε το λόγο κύριε Μακφινά Σκοτ. Λυπούμε που προσήλθαμε καθυστέρηση στην ίδια μου την ακρόαση. Αυτό που ήθελα να πω στην αρχή, ε, καθυστέρησα στην αφήξή μου από το αεροδρόμιο με τον Σερ Πολ Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα στην Κοπενχάγη η διάσκεψη κορυφής για την κρίση του κλίματος. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, η κτηνοτροφία απανταχού έχει με 18% μεγαλύτερο μερίδιο στην έκκληση διοξιδίων του άνθρακος από τις μεταφορές της ίδιας που έχουν 13% υπάρχουν σημαντικά ωφέλη από την κατανάλωση λιγότερων ποσοτήτων κρέατος. Από πέρσι τα Χριστούγεννα δεν έχω φάει κρέας και βρίσκω ότι είναι μια καλή δική μου προσπάθεια. Υπάρχουν πολλές πτυχές. Γεωργία, ανάπτυξη, περιβάλλον. Θα ακούσουμε από τους ε, κοινοβουλευτικούς συναδέλφους μας σήμερα και άλλα σχετικά. Από την Διακυβερνητική Επιτροπή ε, για την Αλλαγή του Κλίματος, Δ. Πατσούρη, και τον κ. Σούτερ που είναι ειδικό εισηγητή των ΗΠΑ, αλλά και από τον ίδιο τον Σερ Πολ Μακάρτνι που ε, έχει, είχε την ιδέα τη ε, Δευτέρα Χωρί Κρέα. Η κτηνοτροφία για κατανάλωση κρέατο, όπω είπα, προκαλεί περισσότερη ε, αναθέρμανση του πλανήτη. Και ε, τώρα, λίγο πριν από τι 10 Δεκεμβρίου, και ως αντιπρόεδρος αρμόδιος για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, σκέφτομαι και εκείνα τα 5 με 7 εκατομμύρια ανθρώπων στις φυλακέ τη Κίνας και στα διάφορα στρατόπεδα ε, που κρατούνται και που δεν λαμβάνουν ποτέ ούτε μία μερίδα κρέατος. Σκέφτομαι και αυτούς. Ε, θα κληθούν τώρα οι κυβερνήσει την επόμενη εβδομάδα να αποφασίσουν για λογαριασμό μα. Αλλά για, από μια άποψη μπορούμε να αποφασίσουμε και εμεί οι ίδιοι και να συμβάλλουμε στην ε, μείωση των συνεπειών τη άλλαγη του κλίματο. Λιγότερο κρέα, λιγότερη αναθέρμανση του πλανήτη. Κύριε και κύριοι, ο Λάινεν. Ευχαριστώ, ε, Έντουαρτ Μακφίναν Σκότ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Μπούσεκ για την εξαιρετική σας ομιλία που κήρυξε την έναρξη των εργασιών μας σήμερα. Λέγομαι Γιώ Λάινεν, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διευθύνω τις ε, συζητήσεις ε, του πάνελ σήμερα. Μετά θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα ακούσουμε τους ε, λόγους του Σερ Πολ και του Ρατσέντα Πατσούρη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε και είναι η κινητήρια δύναμη για την προστασία του κλίματος και έχουμε συμβάλει αποφασιστικά τα τελευταία χρόνια και στην δέσμη μέτρων για την προστασία του κλίματος που ενέκρινε πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε μάλιστα και την αντιπροσωπεία για την Κοπενχάγη ε, με 15 μέλη που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές ομάδες αλλά θα είμαστε και πολύ περισσότεροι διότι το ενδιαφέρον των εκπροσώπων των λαών στην Ευρώπη είναι τέτοιο που θα οδηγήσει τελικά πάνω από 70 ευρωβουλευτές στην Κοπενχάγη και γνωρίζουμε ότι από το Αμερικανικό Κογκρέσο θα έρθουν περίπου 60 από την Βουλή των Αντιπροσώπων και την Γερουσία. Και νομίζω ότι ο ρόλος μας μπορεί να είναι σημαντικός στην Κοπενχάγη. Αν και τα κοινοβούλια δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις αφού αυτές τις διεξάγουν μόνο οι κυβερνήσεις, αλλά εμείς θα είμαστε τα τσοπανόσκυλα που θα παρακολουθούν το τι λένε οι ε, κυβερνήσεις και εάν τηρούν τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Και θα ασκήσουμε και πίεση για να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος για να αναπτυχθεί μια δυναμική τις επόμενες εβδομάδες ώστε και οι κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα από όσα ήδη έχουν υποσχεθεί και όπως είδαμε και στο Μπάλι αλλά και στο Ρίο Δεζανέιρο είδαμε σημαντικά πράγματα που μπορούν να επιτύχουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα κοινοβούλια και ούτω καθεξής. Εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συντάξαμε την έκθεση που ε, ανέφερε προηγουμένως ο Πρόεδρος. Έχουμε και σύστημα ανταλλαγής εκπομπών. Έχουμε και στόχους για την μείωση του διοξιδίου του άνθρακος. Αλλά δεν είναι μόνο η βιομηχανία που πρέπει να αναλάβει δεσμεύσει, είναι και οι μεταφορές με κάθε μορφή τους, όχι μόνο οι οδικές μεταφορές, αλλά και οι εναέρειε μεταφορές, η ναυσιπλοεία, που εκλείουν όλο και περισσότερα αέρια. Και είναι βέβαια και η δασοκομεία και η χρήση των γιών Και θα έρθουμε σε αυτά και θα έλθουμε και στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε τρόφιμα αλλά και παράγουμε τρόφιμα για έναν παγκόσμιο πληθυσμό που μεγαλώνει διαρκώς. Με χαρά θα σας παρουσιάσω τους ομιλητές μας και πρώτος θα είναι ο κύριος Άλαν Ντανκούρ από την ε, Σχολή του Λονδίνου για Υγιεινή και ε, τροπική, ε, θέματα τροπικής υγιεινής. Επίσης οι άλλα μέλη και ο, Κρήτος Αρσέ, Αρσένης που είναι μέλος της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε δημοκρατικές, πολυφωνικές κοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε πολλές απόψεις. Υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή ήδη συμβαίνει και δεν επιτρέπεται να χάσουμε χρόνο για να ε, την αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι αρνούνται την αλλαγή του κλίματος, θεωρούν ότι δεν συμβαίνει τίποτε τέτοιο και αυτοί βέβαια εγείρουν τις φωνές τους και αρνούνται ότι οτιδήποτε έχει σχέση με την παραγωγή του κρέατος μπορεί να επηρεάζει το κλίμα. Όπως είπα, είμαστε open house, είμαστε μια ανοιχτή πολυφωνική κοινωνία και ο καθένας μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του ελεύθερα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο αμέσως στον δόκτορα Άλαν Ντανκούρ για να ακούσουμε τις απόψεις του. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να έρθω να σας μιλήσω. Είναι τιμή μου ε, που είμαι εδώ. Χρειαζόμαστε το φαΐ για να επιβιώσουμε πόσο φαΐ χρειαζόμαστε και τι είδου φαγητό. Ε, ποια θα πρέπει να είναι η μορφή της δίαιτάς μας μέχρι τώρα. Αυτό ήταν ένα ερώτημα που αφορούσε κυρίως ανθρώπους σαν και εμένα. Είμαι διατροφολόγος του δημόσιου τομέα, αλλά και για εκείνου που διαμορφώνουν την πολιτική τη κυβέρνηση είναι θέμα αυτό και εκείνου που δίνουν προσανατολισμό στου καταναλωτέ, τι τρόφιμα χρειάζονται για να προωθούν την υγεία του ο συσχετισμός μεταξύ διαιτός, δίαιτας, διατροφής και υγεία σημαίνει ότι η δημόσια υγεία πρέπει να είναι βασικός, βασικό στοιχείο για να καθορίζονται οι προσανατολισμοί σε εθνικό και σε επίπεδο. Αλλά είναι σαφές τώρα ότι η συζήτηση και η έρευνα για την υγιεινή διατροφή είναι κάτι που χρειάζεται περισσότερους να συμμετέχουν. Επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γινόταν διαχωρισμός μεταξύ πανεπιστημιακών και κυβερνητικών τμήματων και τελικά έτσι ε, δεν υπήρχε συνεργασία μεταξύ των τομέων. Και η κρίση λόγω τη αλλαγή του κλίματο τελικά ε, που αναμένεται θα οδηγήσει σε αλλαγέ και θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλε στρατηγικέ ώστε οι πληθυσμοί να έχουν πρόσβαση και σε υγιεινή και βιώσιμη δίαιτα και διατροφή. Και αυτό θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των ε, προσπαθειών. Ο γεωργικός τομέας ε, συμβάλλει ανάμεσα στο 10 με 12% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σημαντικά ποσοστά προέρχονται από αλλαγές χρήσεως γεών ε, όπως είναι η αποψήλωση των δασών και εκπομπές από τον τομέα θα αυξηθούν κατά μισό της εκατό Δηλαδή 50% περισσότερε εκπομπέ των αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα αυτό μέχρι το 2030. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα γι' αυτό, έτσι δεν είναι. Χρειαζόμαστε φάει, έτσι δεν είναι. Και ο γεωργικό τομέα, δηλαδή οι αγρότε μα δίνουν τα τρόφιμα που τρώμε. Το σικά θέματα θα πρέπει να εξεταστούν. Πόσο φαγητό χρειαζόμαστε, τι είδου τρόφιμα θα πρέπει να παράγουμε και να καταναλώνουμε αν είμαστε σοβαροί για την αποφυγή της αλλαγής του κλίματος. Αυτά είναι σημαντικά θέματα τα οποία συσχετίζουν τη γεωργία με τα τρόφιμα και την υγεία. Και όλα αυτά μαζί με την αλλαγή του κλίματος. Αρχές του έτους μια διεθνή ομάδα επιστημόνων από το συντονισμό τη σχολή του Λονδίνου για τη διατροφή προσπάθησαν να δώσουν κάποια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Εντοπίσαμε ενδεχόμενε στρατηγικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στι κατάλληλε περικοπές εκπομπών των αερίων θερμοκηπίων μέχρι το 2030 στον τομέα των τροφίμων και τη γεωργίας και τότε για πρώτη φορά επίση μπορούμε να αποστατικοποιήσουμε τα αποτελέσματα αυτών των στρατηγικών. Τι συνέπειες θα υπήρχαν για την υγεία των πληθυσμών. Αυτή ήταν ένα πείραμα θεωρητικό σκέψης για να δούμε αν μπορεί να υπάρχει κάποια ωφέλη για την υγεία που προέρχεται από πολιτικέ που ουσιαστικά έχουν σε στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Η δουλειά μα, για εσά που σα ενδιαφέρει, δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα στο Lancet που είναι ιατρικό περιοδικό. Προσπαθήσαμε, ξεκινήσαμε από την υπόθεση ότι οι εκπομπέ αερίου του θερμοκηπίου από τη Γεωργία θα πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθο όπω σε άλλου τομεί, όπω είναι οι μεταφορέ. Ξεκινήσαμε υποθέτοντα ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια των επιλογών σχετικά με το που κάνουμε περικοπέ. Πρέπει να κάνουμε περικοπέ σε όλου του τομεί και βασίσαμε τι εκτιμήσει μα σε στοιχεία για εκπομπέ και στοιχεία για τη διατροφή από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σίγουρα όλοι θα γνωρίζετε ότι ο ΦΑΟ έχει εκτιμήσει ότι η παραγωγή, η κτηνοτροφία ε, ε, συντείνει στα 4, στις 4-5 της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου της Γεωργίας. Οπότε ε, επικεντρωθήκαμε στην κτηνοτροφία. Ίσως μπορούμε να είμαστε πιο αποδοτικοί στη γεωργική παραγωγή προσπαθώντας να μειώσουμε τη σπατάλη και τα απόβλητα αλλά οι στρατηγικέ που επηρεάζουν το μέγεθο τη κτηνοτροφίας ίσω είναι η καλύτερη μέθοδος για να μειωθούν οι εκπομπέ από τον τομέα. Δεν χρειάζεται να τρώμε προϊόντα κτηνοτροφικά όπω είναι το κρέα και το γάλα για την υγεία μα. Σίγουρα στοιχεία διατείνονται ότι κάποια κατανάλωση κρέατος πιθανότατα χρειάζεται τόσο ώστε τα παιδιά που είναι κάτω από 5 ετών να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους ε, όσον αφορά βιταμίνες ε, και κάποια ε, ίχνοστοιχεία. Είναι σαφές ότι η υπερβολική όμως κατανάλωση αυτή των ζωικών προϊόντων συσχετίζεται με προβλήματα υγείας, κακή υγεία κυρίως τους ενήλικες. Παραδείγματος χάρη τα ζωικά προϊόντα συμβάλλουν τα μάλα όσον αφορά τα κορεσμένο ε, λύπη τους ανθρώπους και η κατανάλωση αυτών των κορεσμένων λιπαρών οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Μετά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η μεγάλη κατανάλωση ρηθρού κρέατος και κατεργασμένου κρέατος αυξάνει τον κίνδυνο για κάποια είδη καρκίνων. Η απάντηση στο ερώτημα του κατά πόσο χρειάζεται να τρώμε προϊόντα ζωικά είναι κάτι περίπλοκο να απαντηθεί. Πιθανότατα ναι και σε κάποια στάδια της ζωής μας, αλλά όπως με όλα τα πράγματα πανέτρων άριστον. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη δουλειά μας. Ο γερικό τομέα, επί σειρά ετών προσπαθούσε να βελτιώσει την απόδοση του και να μειώσει τι κομπές αερίων του θερμοκηπίου και έχουν σημειωθεί κάποιε σημαντικέ πρόοδοι. Όμω, οι πρόσφατες εκτιμήσει δείχνουν ότι αυτέ οι στρατηγικές που εφαρμόζονται τώρα όπω η διαχείριση ε, της κοπριάς και σύλληψη ε, του άνθρακου στην ατμόσφαιρα ε, υπολείπονται των στόχων τη Βρετανική κυβερνήσεω για τα θερμοκηπίου και υπολογίζουμε ότι πέραν από τι στρατηγικές που ήδη εφαρμόζονται θα ήταν αναγκαίο να γίνουν περικοπέ όσον αφορά την παραγωγή ζωικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 30% για να καλύψουμε τους στόχους για τα αέρια του θερμοκηπίου στον τομέα της κτηνοτροφίας για το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρωταρχικό στόχο μα και ενδιαφέρον μα δεν ήταν απλώ να εντοπίσουμε ενδεχόμενε στρατηγικέ για να καλύψουμε του στόχου για τα θερμοκηπίου στον τομέα, αλλά ανταυτού να εκτιμήσουμε ποιε συνέπειε θα είχαν αυτέ οι στρατηγικέ επίση επί τη υγεία του πληθυσμού. Γι' αυτό υποθέσαμε ότι η περικοπή 30% στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων θα οδηγούσε σε παρόμοια μείωση στην κατανάλωση των προϊόντων των ζωικών και κυρίως ε, των ε, κεκορεσμένων λιπαρών από ζωικών. Χρησιμοποίησαμε τα στοιχεία που υπάρχουν που συνέδαν την κατανάλωση των κεκορεσμένων λιπαρών με τον κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις ενήλικες καρδιακές παθήσεις είναι το πιο κοινό αίτιο θανάτου στι ανεπτυγμένε χώρε. 7 εκατομμύρια θάνατοι στον κόσμο το χρόνο οφείλονται σε καρδιακέ παθήσει. και η περικοπή 30% στην κατανάλωση των κεκορεσμένων λιπαρών των ζωικών θα οδηγούσε σε ουσιαστική μείωση τη τάξη περίπου του 17% όσον αφορά τον αριθμό των πρώιμων θανάτων από καρδιακέ ασθένειε ε, στους ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή αντιστοιχεί σε 18.000 πρώιμους θανάτους που αποφεύγονται σε ένα χρόνο. Ή περίπου 3% όλων των θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνοψίζοντα λοιπόν, εντοπίσαμε μια στρατηγική για να καλύψουμε του στόχου τη κομπέ αερίων του θερμοκηπίου για τον τομέα τη γεωργία στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή περικοπή της παραγωγής του τομέα της κοινοτροφίας και θεωρήσαμε και εκτιμήσαμε ότι αν οδηγού εφαρμογή στρατηγική σε μείωση τη κατανάλωση των ε, και κορεσμένων λιπαρών από ζωική προέλευση, θα είχαμε βελτίωση τη υγεία του πληθυσμού. Αυτά είναι πολύ καλά μαντάτα. Είναι μια πολιτική που κάνει καλό στο περιβάλλον και κάνει καλό και στη δημόσια υγεία. Είναι μια περίπτωση όπου κερδίζουν όλοι. Εξετάσαμε μόνο μια διασύνδεση διατροφής με υγεία. Ίσως να υπάρχουν και άλλα ωφέλη για την υγεία που συνδέονται με μειωμένη κατανάλωση ζωικών προϊόντων, όπως ε, να έχουμε ε, λιγότερους καρκίνους. Παραδεχόμαστε ότι υπάρχουν αβεβαιότητες όσον αφορά κάποιες, κάποιους υπολογισμούς μας, αλλά απλώς ενδείξεις είναι αυτές για το τι ωφέλη θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε για την υγεία από ομολογικές στρατηγικές που έχουν σαν πρωταρχικό στόχο τη μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου. Βεβαίω υπάρχουν και όροι για όλα αυτά. Οι εκτιμήσει μα βασίζονται μόνο σε στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάποια είδη κτηνοτροφία όπω μικρή κτηνοτροφία για α, στα εγωπρόβατα έχουν μειωμένε εκπομπέ αερίων θερμοκηπίου από ότι η εντατική κτηνοτροφία. Και οι εκτιμήσει μα σχετίζονται με χώρε που κατανόλων μεγάλε ποσότητε ζωικών προϊόντων και για εκατομμύρια ε, ανθρώπους σε φτωχές χώρες τα ζώα είναι σημαντική ε, πηγή διαβίωσης εσόδων. Η πρόταση είναι να μειώσουμε την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων σε χώρες που καταναλώνουν μεγάλα ε, ποσά μεγάλο όγκο τέτοιων προϊόντων. Εμείς δεν προτείνουμε να καταργηθεί η κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Αλλά πόσο ρεαλιστικό είναι κάτι τέτοιο. Πόσο είναι δυνατόν να μετακινήσουμε την κατανάλωση του ε, κοινού, να την αλλάξουμε. Ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο οι άντρες, οι ενήλικες τρώνε πάνω από ένα χιλιόγραμμο κρέατος και ζωικών προϊόντων την εβδομάδα. Προϊόντων κρέατος μάλλον την εβδομάδα. Χρειάζεται τόσο πολύ. Σαφώ δεν χρειάζεται για την υγεία. Και εγώ διατείνομαι ότι η κατανάλωση πολλών ζωικών προϊόντων συνδέεται με πάρα πολύ κακή υγεία, πολύ κακά αποτελέσματα την υγεία. Και αυτό το επίπεδο κατανάλωση κρέατο ε, ε, ξεπερνά τα, τις εθνικές συστάσεις για τη διατροφή. Και εκτιμάται ότι αν τηρηθούν οι εθνικές συστάσεις για τη διατροφή, αυτό ίσως να οδηγήσει σε μείωση για την υγειονομική περίθαλψη στο ύψος των 20 δις ε, λιρών στερλινών στο Ηνωμένο Βασίλειο αρκετές χώρες ήδη ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση της μείωσης της καταναλώσεως ζωικών προϊόντων στους πληθυσμούς τους για το καλό του περιβάλλοντος. Εδώ, στο Βέλγιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι στη Γάνδη ε, αποφάσισαν να μην τρώνε κρέας μία φορά την εβδομάδα. Στη Σουηδία οι κατευθυντήριε γραμμέ για τη διατροφή συστήνουν η κατανάλωση του κρέατος θα πρέπει να μειωθεί λόγω της σύνδεσης αυτής της κατανάλωσης με τα αέρια του και ε, αναφέρεται το ίχνος άνθρακος σε όλα τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης στη Σουηδία. Αυτά είναι γενναία σημαντικότατα βήματα, πρώτα βήματα για την μετώπιση της επικείμενης κλιματολογικής κρίσης. Μεγαλύτερη ευαισθησία του κόστους για το κλίμα όλων των δράσεών μας είναι κάτι πολύ σημαντικό, συμπεριλαμβανομένης τη επιλογή ε, του τι τρώμε. Χρειάζεται να γίνει αμέσως αυτή η ευαισθητοποίηση. Οι κυβερνήσεις και οι καταναλωτές έχουν σκληρέ επιλογέ, δύσκολε επιλογές μπροστά τους, αλλά σίγουρα το να μειωθεί ο ροτάς μας με τα ζωικά προϊόντα ε, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η εισαγωγή. Σε σχέση με την εκστρατεία αυτή για την Δευτέρα χωρίς κρέας θυμάμαι ότι η καθολική μου παιδεία ζητούσε μια Παρασκευή χωρίς Παρασκευή. Αυτό δείχνει ότι εδώ και χιλιάδες χρόνια ξέρουν οι άνθρωποι ότι μία μέρα χωρίς κρέας είναι κάτι θετικό για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχει μια συλλογική λοιπόν σοφία των λαών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ερχόμαστε στα άλλα μέλη του πάνελ. που έχουν στη διάθεσή τους τέσσερα λεπτά και ζητάω από τη Μέρη Μαγκίνες από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σα ευχαριστήσω επίση και για τα τέσσερα λεπτά και για το γεγονό ότι θα με προειδοποιήσετε. Και εγώ καθολική είμαι τώρα που το λέτε. Ίσως λοιπόν η θρησκεία είναι αυτή η οποία παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στις διατροφικές συνήθειες. Μας λέγανε να τρώμε ψάρι την Παρασκευή για να σώσουμε την ψυχή μας. Τώρα μας λένε να μην τρώμε κρέας τη Δευτέρα για να σώσουμε τον πλανήτη. Και νομίζω ότι κανένα από τα δύο αυτά συνθήματα δεν λειτουργεί στην πράξη. Μόνο ένας χορτοφάγος θα ζητούσε να έχουμε μία Δευτέρα χωρίς κρέας. Γιατί έχουμε ψητό συνήθως την Κυριακή στο σπίτι μας και τρώμε τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Δεν τα πετάμε. Αυτό υπομορφή αστείου. Αλλά θέλω να τονίσω τη σημασία αυτής της συζήτησης. Είμαι και μέλος και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, όχι μονάχα Γεωργίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα όλοι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν το λόγο σήμερα ενώπιόν μας να ακούν περισσότερο τις απόψεις ημέν των δε. Πολλές φορές μιλάμε σε διαφορετικούς μονολόγους. Ίσως θα πρέπει να βρούμε μεγαλύτερη απήχηση στα μηνύματά μας μεταξύ μας και θα μάθουμε περισσότερα από τα επιχειρήματα των με και των δε. Ίσως θα μπορούσαμε να τραγουδάμε όλοι το ίδιο τραγούδι. Πρέπει να σας πω ότι η γεωργία είναι ένα μεγάλο κομμάτι του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Σίγουρα η γεωργία και η εκτινοτροφία θα πρέπει να αποτελέσουν τμήμα τη λύσης, αλλά δεν είναι η μόνη λύση. Αν εξετάσουμε την ευρωπαϊκή γεωργία, έχει καταβάλει τεράστιε προσπάθειε, επιτυχεί προσπάθειες για να μειώσει τι εκπομπές αριών θερμοκηπίου. Οι γεωργοί, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της κτηνοτροφίας και του φυσικού περιβάλλοντος, αυτοί θα έπρεπε να είναι παρόντες στη σημερινή συζήτηση και ακόμα και στο πάνελ για να δώσουν την άποψή τους. Αλλά έχουμε μειώσει εκπομπές από την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ξέρουμε με ποιο τρόπο θα το κάνουμε. Και η έρευνα μας κατευθύνει προς την κατεύθυνση περισσότερων βελτιώσεων και οι γεωργοί θα ήθελαν να ξέρουν ποιες είναι αυτές οι προτάσεις. Μας έδωσε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία ο τελευταίο ομιλητή δεν είπε να αφαιρέσουμε τελείως το κρέας από την ανθρώπινη διατροφή. Είναι πολύ μέσα σε αυτή την ε, αίθουσα και δύο ή τρεις από τους κύριους ομιλητές ζήτησαν να αφαιρεθεί τελείως το κρέας από την διαιτά μας. Εγώ διαφωνώ με αυτή την πρόταση. Διαφωνώ από πολλούς, για πολλούς λόγους. Δεν είμαι διαιτολόγος. Είμαι μητέρα παιδιών όμως και ξέρω ότι πρέπει εγώ να φροντίζω το τι τρώει ο κόσμος στην οικογένειά μου. Νομίζω ότι μια μετριοπαθής αντιμετώπιση, μια αντιμετώπιση πανμέτρων άριστον είναι το καλύτερο. Εγώ χαίρομαι να έχουμε κρέας πολλές φορές και δεν θέλω να πείσω κανένα να ακολουθήσει δικές μου διατροφικέ συνήθειες να τρώμε γαλοπούλα, πραγματικά να τρώμε ε, πόριτ το πρωί κάθε μέρα. Αυτό είναι θέμα του καθενός που μπορεί να το διαλέξει μόνος του. Ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνται οι εκπομπέ από τη γεωργία, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθούν να αυξάνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντική η κτηνοτροφία στον αναπτυσσόμενο χώρο και ανησυχώ ότι το μήνυμα το οποίο θα δώσουμε εμεί μπορεί να έχει αρνητικέ επιπτώσει στον αναπτυσσόμενο κόσμο και θα επηρεάσει το γεγονό ότι για αυτού η κτηνοτροφία είναι σημαντική όχι μόνο για τη διατροφή αλλά και σαν μέσο εργασίας και μεταφοράς ο αναπτυσσόμενος χώρος και οι αναδυόμενες οικονομίες θέλουν να μιμηθούν τα δικά μας διατροφικά πρότυπα. Δεν θέλουμε να είναι υπερβολικοί, υπερβολικοί καταναλωτές οποιοδήποτε προϊόντος, ούτε να μιμηθούν τις κακές μας συνήθειες. Αλλά μην δίνετε την εντύπωση ότι αν γίνουμε όλοι χορτοφάγοι θα έχουμε μικρότερο πρόβλημα σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής. Σήμερα το πρωί μπήκα σε αυτή την αίθουσα και πολλοί από εσά καταλάβατε ότι ήταν πολύ ζεστή η αίθουσα και αυτό πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Είναι πολλοί τρόποι με τους οποίους εμείς διδάσκουμε τους άλλους τι πρέπει να κάνουν αλλά δεν ακολουθούμε αυτό το παράδειγμα. Δάσκαλε που δίδασκε. Είναι πολύ απλό να μειώσουμε τη θερμοκρασία μια αίθουσα. Μου είπαν όμω ότι το σύστημα δεν το επιτρέπει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τη γεωργία. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπο αντιμετώπιση τη γεωργία. Έχω ακόμα χρόνο. Λίγο χρόνο ακόμα, μόνο θέλω. Έχει αλλάξει πάρα πολύ λοιπόν η λειτουργία της γεωργίας και θα εξακολουθήσει να αλλάζει, αλλά εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι πρέπει να υπάρξει και κτηνοτροφία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να γίνει καλύτερα αυτή η κτηνοτροφία και την έχουμε βελτιώσει ήδη. Αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται λοιπόν την ε, γη δεν θα πρέπει να βρεθούν εκτός συζήτησης. Δεν πρέπει οι κτηνοτρόφοι να προσβληθούν από το μήνυμα της σημερινής μας συζήτησης. Θα πρέπει να τους συμπεριλάβουμε στη συζήτηση για να μπορούμε να έχουμε από κοινού όλη πρόοδο. Ευχαριστώ, Μέρι Μαγκίνες, από την Επιτροπή Γεωργίας. Η γεωργία δεν είναι το πρόβλημα, είναι τμήμα μοναχά του προβλήματος, αλλά υπάρχει και η θέληση να είσαστε τμήμα της λύσης. Τρώτε ψητό την Κυριακή και τη Δευτέρα τα υπόλοιπα. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τι γίνεται στην Ελλάδα. Ο Κρήτορα Ρασένης από την Επιτροπή και, και από την Επιτροπή Περιβάλλον. Ε, για την Επιτροπή Ανάπτυξη, συγγνώμη. We do not know enough about this anthropogenic climate change. Δεν γνωρίζουμε αρκετά για τους ανθρωπογενείς παράγοντες της αλλαγής του κλίματος. Όταν έγινε Ευρωβουλευτής αναζήτησα τρόπους ε, για να συμβάλλω στην αντιμετώπιση αυτών των ε, απειλών. Και καταλαβαίνω ότι δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί ο, ο πλανήτης και το κλίμα του και πρέπει να τα καταλάβουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουμε αντιμετωπίσει παρόμοιες απειλές στην ανθρωπότητα και πριν, όπως τον ψυχρό πόλεμο και την πυρηνική απειλή όπου είχαμε ή τον Ρίγκαν ή τον Γκορμπατσόφ ή κάποιον άλλο που θα πατούσε ένα κουμπί για να κάνει το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Τώρα η απειλή είναι διαφορετική. Ο καθένας από εμά που πατάει το κουμπί του διακόπτη για να ανάψει το φως ή να το κλείσει ή για να βάλει μπρο στον κινητήρα του αυτοκινήτου του ή ε, στο μηχάνημα του εργοστασίου. Όλα αυτά αποτελούν απειλή. Δεν γνωρίζουμε όμω όλε τι διασυνδέσει των παραγόντων αυτών στην φύση. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πόσε από όλε αυτέ τι δραστηριότητε μα επιταχύνουν τι αλλαγέ του κλίματο. Για μένα η συζήτηση είναι σημαντική, διότι προσθέτει μία παράμετρο ακόμη στην συζήτηση, ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε ακόμα υπόψη μας. Η ΦΑΟ υπολόγισε ότι η συμβολή των, ε, ε της κτηνοτροφίας είναι περίπου 18%. Αλλά από το World Watching Institute ανεβάζουν τη συμβολή αυτή στο 51% γιατί θεωρεί ότι η ΦΑΟ χρησιμοποίησε διαφορετικά δεδομένα. Ίσως είναι υπερβολή, αλλά ε, πάντως αυτό που μας λέει είναι ότι η κτηνοτροφία συμβάλλει ε, σημαντικά στην αλλαγή του κλίματος. Και βέβαια η κατανάλωση ενέργεια βέβαια ε, για την κτηνοτροφία περιλαμβάνεται στου υπολογισμού αυτού. Εμεί λοιπόν καταναλώνουμε τώρα τα προϊόντα τη κτηνοτροφία. Και όπω είπε η κυρία Μαγκίνε, μειώνεται η γεωργία στην Ευρώπη συνολικά, αλλά η κατανάλωση προϊόντων κτηνοτροφίας αυξάνεται σημαντικά. Είτε λοιπόν ε, καταναλώνουμε δικά μας, τα προϊόντα της δική μας κτηνοτροφίας, είτε τα εισάγουμε, πάντως καταναλώνουμε όλο και περισσότερο κάθε χρόνο. Εμείς λοιπόν, οι Ευρωπαίοι, είμαστε αυτοί που πληρώνουμε ώστε σε άλλα μέρη του πλανήτη να καταστρέφονται τα, τα δάση για να γίνουν βοσκοτόπια, για να βοσκήσουν ζώα όπου τελικά εμείς θα καταναλώσουμε τα προϊόντα της κτηνοτροφίας αυτής. Άρα είναι μια ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι. Εγώ προερχόμενος από χώρα της Μεσογείου, η ε, λύση που βρίσκω εγώ είναι οι τοπικές μας δίαιτες, που δεν περιλάμβανε ασφαλώς την κατανάλωση κρέατος καθημερινά. Ε, ε, τώρα βέβαια ναι. Είναι όμως πρόσφατη εξέλιξη αυτή και εντάσσεται μέσα στον καταναλωτισμό μας. Η πρότασή μου λοιπόν ε, για μια βιώσιμη παραγωγή τροφίμων θα ήταν να, ξανα, να επιστρέψουμε ξανά στις ε, ρίζες μας, στις παραδόσεις μας για τη διατροφή μας που είναι και πιο ενταγμένη, πιο ε, συναρμοσμένη στις ικανότητες των ντόπιων κοινωνιών να παράγουν αυτά που χρειάζονται για την καταναλώτησή τους. Ευχαριστώ πολύ, Κρήτονα. Μεσογειακή δίαιτα είναι παγκοσμίω φημισμένη. Μπορεί να δει κανείς και, ποια, και ποιες ασθένειες απουσιάζουν όταν τρώει κανείς τούτο τρόπος. Έχουμε 50 λεπτά χρόνο συζητήσεως στην Ολομέλεια. Στο, εδώ στο κοινοβούλιο, στην αίθουσα, είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες. Μπορείτε να μιλήσετε όποια γλώσσα θέλετε, δηλαδή την ε, μητρική σας γλώσσα. Έχουμε μια διαδικασία που τη λέμε ε, διεθνώς catch the eye, δηλαδή όποιος ε, σηκώσει το χέρι του και τον δύο πρόεδρος θα του δώσει το λόγο. Θα προτείνω όμως ένα-ενάμιση λεπτό για τον καθένα σας δεν είναι πολλοί, αλλά μπορείτε να εκφράσετε μία ή δύο ιδέε και έτσι να έχετε τη δυνατότητα να συμβάλλετε στη συζήτηση. Ποιο επιθυμεί να λάβει το λόγο. Βλέπω ότι τα μέλη μας ενδιαφέρονται πολύ. Έχετε το λόγο παρακαλώ κύριε εσείς. Παρακαλούμε να αυτοσυστηθείτε. Να πείτε το όνομά σας και από πού προέρχεστε. Ρόλφ λέγομαι. Είμαι πρόεδρος της ε, Ένωσης των ε, Γεωργών στην Ευρώπη. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμβάλλω σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία πρέπει να αναφερθούν. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τους ε, υπολογισμούς για τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίου δεν υπάρχει λήψη υπόψη του γεγονότος ότι η παραγωγή, η κτηνοτροφική παραγωγή γίνεται σε, σε λιμόνες, σε λιβάδια που είναι χώρος απόθεσης ε, διοξιδίου του άνθρακος. Απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακος οι λιμόνες. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να καταλογιστεί μέσα στα πλαίσια της συνολικής ισορροπίας του διοξιδίου του άνθρακος. Αν το δείτε με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ χαμηλότερες οι εκπομπές από την κτηνοτροφία είναι πραγματικά μικρότερες κατά 30 50% από τα στοιχεία τα οποία παρουσιαστήκαν. Επίσης, είπατε ότι χρησιμοποιείτε, κάποιος ομιλητής είπε ότι χρησιμοποιεί στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά 60% της έκτασης του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρρώσιμες καλλιέργειες παρά μόνο για λιμόνες και για ε, ε χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αν λοιπόν πάψουμε να έχουμε κτηνοτροφία δεν θα είμαστε σε θέση να διατρέφουμε όλο τον κόσμο. Το 60% αυτό το ποσοστό είναι ακόμα πιο ψηλό σε άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία από την οποία προέρχομαι. 80% της έκτασης της Ιρλανδίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλλιέργειες. Επομένως χωρίς παραγωγή κτηνοτροφική και γαλακτοκομική παραγωγή δεν θα μπορούσε να υπάρχει καμία αγροτική δραστηριότητα και διατροφή. Επίσης η παρουσίαση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι αν περάσουμε από μια δίαιτα που βασίζεται στο κρέας σε μια <clears throat> δίαιτα που βασίζεται σε χορτοφαγία αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες εκπομπές γιατί όταν ε, οργώνουμε τη γη απελευθερώνουμε ποσότητες διοξιδίου του άνθρακος ενώ όταν έχουμε απλώς χορτολιβαδικές εκτάσεις έχουμε αποθετήρια διοξιδίου του άνθρακος. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συμβολή σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιέρ Σεβαλή είναι το όνομά μου πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας για τα Βοηδή της Γαλλίας, πρόεδρος της ομάδας ε, του Βοήου Κρέατο στην Κόπα Κοζεκά. Ευχαριστώ Πρόεδρε που οργανώσετε αυτή τη συζήτηση για την ε, θέρμανση της ατμόσφαιρας και για το κλίμα παραμονής Κοπεχάγη. Η ποιότητα των ε, παρεμβάσεων που προηγήθηκαν ήταν πάρα πολύ καλή. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που υπόθηκαν και σήμερα εδώ, σε αυτό το βήμα που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να κάνουμε τη διαφορά, τη διάκριση μεταξύ Ευρώπη και των, μεγάλων, των άλλων μεγάλων υπήρων παραγωγή βοήου κρέατο. Στην Ευρώπη παράγουμε βόηο κρέα πάνω σε εκτάσει όπου η διατροφή των βοηδών γίνεται κατά 80% από τα λιβάδια, από τους λιμόνες. Είναι λιμόνες εκεί και είναι πραγματικά παγίδε άνθρακο οι λιμόνε. Απορροφούν τον άνθρακα. Και αν κάνουμε σύγκριση σε παγκόσμιο επίπεδο τη κατανάλωση βοηού κρέατο, βλέπουμε ότι στη Γαλλία καταναλώνουμε δύο ε, μπριζόλε την εβδομάδα. Μα μένουν ακόμα πολλέ ημέρε, δηλαδή πέντε ημέρε για να καταναλώσουμε κάτι άλλο. Και όταν το μέσο όρο ευρωπαϊκή καταναλώσεω βοηού κρέατο κατά κάτοικο είναι 15 κιλά, είναι 70 κιλά στην Νότια Αμερική και 50 κιλά στι ΗΠΑ. Είναι πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση των αερίων του θερμοκηπίου και της διατροφής και να δούμε τι γίνεται στην κατάσταση που κρατεί στην Ευρώπη και μην τα αναμίξουμε αυτά με την παγκόσμια κατάσταση. Έχουμε εκτατική κτηνοτροφία. Ε, χωροταξία ακολουθούμε στην Ευρώπη, διατηρήσεω των ειδών τα είδη τα οποία ζουν στην Ιρλανδία ή στις περιοχές της Γαλλίας, τους λιμόνες της Νορμανδίας, όπου η παραγωγή γάλακτος και βουίου κρέατος είναι κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ισορροπία τη χωροταξική και την ισορροπία της κοινωνίας. Συνεπώς, ας μην αναμειγνύουμε την ευρωπαϊκή κατάσταση με την κατάσταση που επικρατεί στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεβαλιέ. Επόμενος, Βιτόριο Πρόντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Και εδώ παίζονται πολύ σημαντικές ισορροπίες. Το έδαφος έχει περιεχόμενο άνθρακος που είναι το διπλάσιο από αυτό στην ατμόσφαιρα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα να ε, κρατήσουμε ε, την κατάσταση ως έχει το πρόβλημα της κτηνοτροφίας η κτηνοτροφία βασίζεται σε προϊόντα της αρρώσιμης γης όμως στον αραβόσιτο Φερρυπίν 8 χιλιόγραμμα αραβοσίτου χρειάζονται για παραγωγή ενός χιλιογράμμου κρέατος άρα θα μπορούσαμε να διωτηθούμε τι χρειάζεται για τις ίδιες πρωτεΐνες υπό τη μορφή γάλακτος. Το πρόβλημα είναι να δούμε συνολικά το πρόβλημα, να βρούμε σωστή ισορροπία, βέλτιστη ισορροπία για την χρήση των αρρωσίμων γεών, δηλαδή χρήση για κτηνοτροφία και χρήση για την παραγωγή ε, τροφίμων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Κάρολαϊν Λούκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι μέλο των Πρασίνων στο Ηνωμένο Βασίλειο και χαιρετήσω ιδιαίτερα τη σημερινή συζήτηση. Πολλοί από εμά προσπαθούν να θέσουμε αυτό το θέμα των εκπομπών από την κτηνοτροφία στη μέση διάταξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χαίρομαι που σήμερα επιτέλου λαμβάνετε στα σοβαρά αυτό το θέμα. Έχω μία ερώτηση και ένα σχόλιο να σα υποβάλω. Το ερώτημα είναι για τον πρώτο ομιλητή από το Σχολείο Δημόσιας Υγείας του Λονδίνου. Είπε ότι τα παιδιά χρειάζεται να έχουν κρέας στην παιδική ηλικία για να έχουν μια ισορροπημένη ανάπτυξη. Δεν ξέρω ποια είναι τα επιστημονικά πορίσματα που οδηγούν σε κάτι τέτοιο. Είναι πιο δύσκολο να έχει κανεί πιο ισορροπημένη δίαιτα χωρί κρέα, αλλά πιστεύω ότι είναι δυνατόν να το επιτύχει αυτό και χωρί κρέα. Δεν ξέρω ποιε επιστημονικέ μελέτε οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα το οποίο αναφέρατε. Χρησιμοποίησατε επίση μια άλλη φράση. Είπατε μια λύση win-win που κερδίζουν όλοι. Ότι αυτό βοηθάει το κλίμα και βοηθάει και την ανθρώπινη υγεία. Εγώ θα ήθελα μια κατάσταση που είναι win-win-win-win, που κερδίζουμε όλοι και ξανακερδίζουμε όλοι. Θα είναι καλό και για την ευζοία των ζώων, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα σήμερα, γιατί ξέρουμε ότι η εντατική παραγωγή κρέατος έχει αρνητικό αντίκτυπο στα ζώα και επομένως Θέλω να τονίσω ότι ο προηγούμενος ομιλητής μίλησε για το ποσοστό μετατροπής των πρωτεϊνών από τον αραβόστο στο κρέας. Αν θέλουμε να διαθρέψουμε ένα αυξανόμενο πληθυσμό σε επόμενες δεκαετίες, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να διαθρέψουμε ένα τέτοιο πληθυσμό που αυξάνει με τα διατροφικά τρόφιμα τη Δύση. Πρέπει να έχουμε μια δίαιτα η οποία θα έχει λιγότερο κρέας, γιατί αλλιώ αυτό σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ σπάταλοι σε ό,τι, σε ό,τι αφορά τη Χριστό Δημητριακό για την παγκόσμια διατροφή. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Oui, bonjour, je suis parlementaire belge, Είμαι Βελγίδα οικολόγος βουλευτής θα ήθελα να προτείνω το εξής, ότι από τη συζήτηση αυτή θα πρέπει να αποκομίσουμε και μια μεγαλύτερη σκέψη σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ε, καλλιέργειας σιτηρών και της ε, κτηνοτροφίας. Η κτηνοτροφία εξάλλου μας δίνει λιπάσματα για τη γεωργία, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα ζώα θα πρέπει να διατρέφονται από χόρτο και με τον τρόπο αυτό είναι πιο καλό το αποτέλεσμα και για την υγεία μας, δεν υπάρχουν υπερβολικά λύπη στα ζώα. Είναι σημαντική λοιπόν η διατροφή και των ζώων. Το ερώτημα επομένω που πρέπει να θέσουμε είναι αν η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική ενθαρρύνει την εκτατική εκτροφή των ζώων και όχι την εντατική εκτροφή και τις ε, μορφές εκτροφής που βασίζονται σε εισαγόμενες φυσικές, φυτικές πρωτεΐνες ή αραβόστο και που οδηγούν στο να έχει η Ευρώπη ένα μεγάλο οικολογικό χρέος μέσα σε εισαγωγικά έναντι άλλων χωρών. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε ότι μια εκτροφή που βασίζεται στο έδαφος, αυτό θα πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να υποστηρίξει η αγροτική μας πολιτική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχει το λόγο κυρία μου. Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Γεωργών είμαι έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα απευθυνόμενοι στον εκπρόσωπο του London School of Hygiene για το περιεχόμενο σε κορασμένα λιπαρά που αναφερθήκατε όσον αφορά την κτηνοτροφία και τα ζωικά προϊόντα. Δεν υπάρχει κανεί σε αυτή την αίθουσα που θα διαφωνούσε μαζί σα αν λέγαμε ότι η κατανάλωση των Hamburger κάθε μέρα είναι κάτι κακό για την υγεία σου. Αλλά καμιά φορά είναι και η κατεργασία των προϊόντων που παίζει σημασία. Κάτι που αφορά την παραγωγή και όχι, και όχι σε επίπεδο Εκμετάλλευση που υπάρχει το πρόβλημα. Έχετε κάποιες πληροφορίες γενικά όλοι σας το πώ αλλαγή διατροφή των ζώων της συνοτροφία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση εκπομπή μεθανίου παραδείγματο χάρη σε επίπεδο των εκμεταλλεύσεων. Εσείς έχετε το λόγο. Hello, my name is Sebastian Tosh. I'm from... Sebastian Tosh, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χορτοφάγων. ακούστηκε κάποια δήλωση ότι πρέπει να τρώει κανείς κρέας σε κάποια φάση της ζωής του. Θα ήθελα να πω και εγώ κάτι. Υπάρχει η Αμερικανική Διατολογική Ένωση, η μεγαλύτερη ένωση διατροφολόγων και διατολόγων, και έχουν, εκπονούν κάθε χρόνο έγγραφο για τη χορτοφαγία και λένε ότι ακόμα και η καλή κατανάλωση η χορτοφαγική ε, κατά όλη τη διάρκεια της ζωής σου ε, μπορεί να είναι εφικτή και κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, εγκυμοσύνης λοιπά Ακόμα και αν δεν φας ποτέ στη ζωή σου ζωικά προϊόντα μπορείς να ζήσεις ε, πολύ υγιεινά. Ευχαριστώ. Κούν Μπούκαρτ um, από την ε, ε, ε, Ένωση μεταποίηση Σόγια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές για να περάσουν από ένα πρότυπο που βασίζεται στην κατανάλωση ζωικών προϊόντων σε ένα πιο χορτοφαγικό πλαίσιο. Εμείς ως παραμεταποιητές σόγια στην Ευρώπη προτείνουμε και νέες λύσεις, παραδείγματος χάρη γάλα από σόγια, για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των καταναλωτών. Είναι πολύ καλό σε ό,τι αφορά τη γεύση, χαμηλή περιεκτικότητα σε χολυστερίνη και σε κεκορεσμένα λίπη, πολύ υγιεινή λέει, πολύ υγιεινά προϊόντα λοιπόν το γάλα από σόγια και είναι μια πρακτική λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα. Επίσης θεωρούμε ότι τα προβλήματά μας έχουν και μικρότερο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την εκπομπή διοξίδου του άνθρακος πέντε φορές λιγότερο εκπομπές διοξιδίου του άνθρακο σε ό,τι αφορά τις ε, εκπομπές από προϊόντα σόγιας και ένα παράγοντα δύο σε ό,τι αφορά το κρέας. Όλα αυτά, το αντίστοιχο του κρέατος, όλα αυτά λοιπόν μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε λιγότερη κατανάλωση ύδατος, λιγότερες εκπομπές. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να έχουμε πρακτικές λύσεις σε ό,τι αφορά την διατροφή των καταναλωτών και η απάντηση μπορώ να πω ότι ήδη τα προϊόντα αυτά βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Όταν σκεφτόσαστε λοιπόν για τις εναλλακτικές αυτές λύσεις μέσα στην νομοθεσία, τότε μια οργάνωση σαν τη δικιά μας μπορεί να εξασφαλίσει μια λύση εάν υπάρξει μια μη διακριτική αντιμετώπιση των προϊόντων που έρχονται από σόγια σε ό,τι αφορά τη διατροφική αξία και τη μείωση των εκπομπών. Πέρα σύμβουλος στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ό,τι χρειαζόμαστε, το μόνο χρειαζόμαστε είναι φαγητό. Φαγητό, αλλά καλό φαγητό. Μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι ένα γεύμα το 2030, όταν εγώ θα είμαι 74 ετών. Θα είναι μόνο φλούδια, μόνο χάπια το 2030. Ίσως να συνθέτει και ένα τραγούδι ο Πολ Μακάρτνη. Λοιπόν, ως συνήθως ο κίνδυνος να παίζω σε κάποιο έργο αισθάνομαι. Είναι σαν να βρισκόμαστε στο τρελοκομείο. Έχουμε, ε, βλέπουμε τη αφάξη της δημοκρασίας που αναφέρεται. Γιατί είχε ζεσταθεί το μεσαίωνα ο κόσμος και ήταν πιο ζεστός σε συγκρίση με σήμερα. Εδώ και 2.000 χρόνια ήταν πιο θερμό, κατά τη διάρκεια τη θερμή περίοδου τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που στη Σκωτία ακόμα παρήγαγαν ε, κρασί. Δεν έχει, ε, την τελευταία δεκαετία δεν έχει ζεσταθεί ο πλανήτη. Κοιτάξτε το, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί την αλλαγή του κλίματο και την αύξηση τη θερμοκρασία για να δικαιολογήσει την ύπαρξή τη. Και ο Καϊκομήρη, ο Πολ Μακάρνι, ξεγελάστηκε. Αυτό που είπατε εσεί, Πρόεδρε, στην αρχή. Είπατε ότι αυτοί που είναι διστακτικοί, σκεπτικιστέ όσον αφορά την αλλαγή του κλίματο είναι αρνητέ. Είστε Γερμανό και ξέρετε τι σημαίνει αυτό ο όρο και θα πρέπει να μα αποκαλείτε σκεπτικιστέ. Γιατί αυτό μα Ο κ. Μακμίλαν Σκοτ είπε ότι πήγε στο αεροδρόμιο να μαζέψει τον κύριο Μακάρτνεϊ. Λοιπόν, δεν πράττει τα όσα κηρύσσει. Εμείς στο κόμμα ανεξαρτησίας ε, ετοιμάζουμε μπάρμπεκι απ' έξω ψισταριά ο τίτλος μας είναι «Το μόνο που χρειάζεσαι είναι κρέας». All you need is meat και σερβίρουμε κρέας στις 12 το μεσημέρι. Απολαύστε το φαγητό σας και ελπίζω να μην έχει συνέπειες για εσάς, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Κυρία μου. Ε, Joyce De Silva από την ε, Γεωργία με, με συμπόνια. Πρέπει να σας πω ότι οι στατιστικές του ΦΑΟ δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα διπλασιαστεί ο αριθμός των ζώων που εκτρέφονται στον κόσμο μέχρι το 2005. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Ένα τρίτο όλων των δημητριακών στον κόσμο πηγαίνουν για ζωοτροφές. 94% της σόγιας η οποία καλλιεργείται πηγαίνει για ζωοτροφές επίσης. Ενώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τα και όταν χρησιμοποιούμε τα δημητριακά για βιοκαύσιμα, αυτό σημαίνει ακόμα λιγότερα τρόφιμα για τους ανθρώπους. Ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων πεινάνε κάθε βράδυ όταν εμείς δίνουμε τα δημητριακά στα κοτόπουλα, στα γουρούνια, στα βόηδη για να έχουν περισσότερο κρέας, περισσότερα αυγά κτλ. Και επίσης θέλουμε και τα αυτοκίνητά μας να τα τροφοδοτούμε με βιοκαύσιμα. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα την Κάρολιν Λούκα σε σχέση με αυτό που είπε για την ευζοία των ζώων γιατί πράγματι ο κύριος μου κάνει λάθος. Δύο τρίτα των ζώων που χρησιμοποιούν για την κτηνοτροφία βρίσκονται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν έχουν σαν προτεραιότητα την ευζοία των ζώων, ζουν σε άθλιες κατάσταση αυτά τα ζώα και δεν μπορούν να ζήσουν σε φυσικό, με φυσικό τρόπο. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μία κατάσταση win-win παρά μόνο αν εκτρέχουμε τα ζώα με ανθρώπινο τρόπο σε χορτολιβαδικές εκτάσεις και σταματήσουμε την, την ε, εντατική κτηνοτροφία, τα ζώα αυτά θα είναι πιο ευτυχισμένα. Επόμενο Επόμενος ομιλητής. Περπατάει πίσω από εκείνον που ετοιμάζει την ψισταριά, δεν μπορώ το στο λόγο. Θέλετε να φάτε το... την πριζόλα σας, Chris Chris, θα ήθελες να πάρεις το λόγο. Γιατί είσαι ο τελευταίος πριν δώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ και μετά πάμε στο διάλειμμα του καφέ. Βλέπεις πόσο ελκυστική είναι η ψησταριά ε, για το φίλο μας. Ξέχασε ότι θα πάρει το λόγο. Αλλά τώρα η παρέμβασή του σίγουρα δεν θα ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση της κρατοφαγής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον συνάδελφο, τον Πολ Νάτα, από την περιοχή μου, που έμεινε για να μπορέσω να τον προσβάλλω. Καταρχά να πω ότι είναι κάποια στοιχεία τη συζήτηση που είναι τεχνητά, είτε είσαι χορτοφάγο ή σαρκοφάγο. Κοιτάξτε τώρα, οι περισσότεροι από εμά είμαστε πανφάγα και υπάρχουν λόγοι υγεία που θα πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση κρέατο στον κόσμο και υπάρχουν και περιβαλλοντικοί λόγοι για το, προς την ίδια κατεύθυνση. Χρειάζεται ισορροπία σε όλα. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη για το εκπαιδευτικό σύστημα στη βορειοδυτική Αγγλία που παράγει κάποιον που πιστεύει ότι το ότι επειδή είχαμε ζεστή χρονιά το 98 δεν δείχνει ότι έχει αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη και λυπάμαι ότι κανένας δεν τον δίδαξε τον νόμο του όρου. και ζητώ συγγνώμη επίσης διότι οι πόλεις που εκπροσωπώ και ο Πολ Νάτερ, το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ πολλές φορές διαπίστωνα ότι υπήρχαν τεράστιε διαφορέ από, κάθε από μια περιοχή στην άλλη όσον αφορά το προσδόκιμο ζωή. Και ένα κομμάτι των, ε, του αιτίου είναι και η διατροφή. Και οι φτωχοί τρώνε πράγματα, έχουν άλλη διατροφή. Και τα λιπαρά συμβάλλουν ιδιαίτερα στη διατροφή τους και αυτό οδηγεί σε καρδιακές ασθένειες και μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Αυτό είναι κάτι που είναι σοβαρό. Θα πρέπει το θέμα τη διατροφής διατροφή να εξεταστεί. Οι φτωχότεροι στο Λίβερπουλ και στο Μάντσεστερ έχουν δικαίωμα να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωή, όπω και ε, τη μεσαία τάξεω. Και λυπούμε που το UKIP πιστεύει ότι όλα αυτά είναι απλώ ένα αστείο, μεγάλο αστείο. Yeah, Σας ευχαριστώ. Οι παρεμβάσει ήταν όλε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε. Μπορούν τώρα τα μέλη ε, του πάνελ να, να σχολιάσουν. Κρήτον θέλετε εσείς να λάβετε πρώτο το λόγο. Θέλω μόνο να προσθέσω ότι υπάρχει και το θέμα του πώς εκτρέφονται τα ζώα και αυτό είναι σημαντικό και σημαντικό θέμα και πολιτιστικά. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά στην νοοτροπία μας γιατί πολλά που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την ε, νοοτροπία μας, αυτόν τον πολιτισμό μας είναι και αυτά τα οποία είναι συνυπεύθυνα για την, ε, για την ε, έκκληση του διοξιδίου και την αλλαγή του κλίματος. Ορισμένες παρεμβάσεις ακούσαμε για τον τρόπο που ε, παράγονται τα τρόφιμα. Ναι, εγώ δεν θα είμαι τόσο σύντομη και ζητώ να δείξετε κατανόηση. Οι παρεμβάσεις δείχνουν πόσο ποικίλουν οι απόψεις ο Chris Evans νομίζω ότι τα είπε σωστά. Συμφωνώ με αυτά που είπες ότι οι φτωχοί ε, διατρέφονται και χειρότερα και ότι το θέμα της αλλαγής του κλίματος είναι περισσότερο θέμα των ε, μεσαίων τάξεων. Μακάρι να προερχόταν η συζήτηση αυτή από αυτούς που πλήττονται και περισσότερο. Αλλά πάντως Υπάρχουν διαφορέ αυτέ αποκλήσεων και αν είναι έτσι μονομερή τα θέματα δεν πρόκειται να ε, προωθηθούν. Εγώ προέρχομαι από τη Γεωργία. Για θέματα ευημερία των ζώων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τι πιο αυστηρέ διατάξει σε όλα τα συστήματα παραγωγή δεν κάνει τίποτα ωστόσο, για παράδειγμα, στο επίπεδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στη Γενέβη, καθώ τώρα μιλούμε, προχωρούν με ακόμα περισσότερη απελευθέρωση τη αγορά. Για όλου εμά που, που είμαστε εύποροι, είναι ότι δεν πληρώνουμε υπερβολικά για τα τρόφιμα που αγοράζουμε, δεν, τους, δεν ανταμείβουμε αρκετά του γεωργού για την υπηρεσία που προσφέρουν στο κοινό. Και μέχρι, αν εφόσον δεν το κάνουμε αυτό, σπρώχνουμε τους γεωργούς να παράγουν όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες τους. Αυτά εμάς μας ενοχλούν. Εμείς πληρώνουμε για να εκτρέφεται κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να μας αγοράσει και να μας φάει όλους. Αλλά το μήνυμα είναι όταν θα φύγει από εδώ είναι για μας τους εκλεγμένους πολιτικούς εμείς θα μείνει να, να ε, τηρήσουμε τις υποσχέσεις, τα υπεσχημένα. Εγώ θεωρώ και κυρίως για τα βοσκοτόπια, μία πολύ νεαρά κυρία νομίζω κυρία Φίλτς Πάτρικ που ρώτησε σχετικά με την έρευνα. Ναι, γίνεται πολύ έρευνα και στην Ευρώπη αλλά και στην Αυστραλία για το τι πρέπει να τρώνε τα μυρικαστικά αλλά και αυτά τα πολιτικά για το ποιο τρώει κρέα, το ποιο τρώει ε, μόνο φυτοφαγικά, το ποιο δεν τρώει καθόλου προϊόντα ε, ζώων. Ναι, και εγώ είμαι μητέρα και ε, έχω ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Thank you. Ευχαριστώ. Ο Δόκτωρ Νταγκούρ για δύο-τρία λεπτά, αν μπορείτε να σχολιάσετε κι εσείς. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχει προκαλέσει τόση πολλή συζήτηση το θέμα αυτό και ο καθένα έχει άποψη για τα θέματα αυτά, γιατί τα θέματα τα διατροφικά είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλου μα. Μα νοιάζει το τι τρώμε. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε περισσότερο για τη διατροφή μα και πρέπει να σκεφτούμε και για τι επιπτώσει στο περιβάλλον τη διατροφή μα. Θέλω να σταθώ σε μερικά σημεία μονάχα που αναφέρθηκαν και να δώσω μια απάντηση. Πρώτον, το σημαντικό θέμα για, τις, για τους λιμόνες και την κτηνοτροφία. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πιο σημαντικό από όλα όμως είναι η, ποια είναι η κλίμακα της ε, κτηνοτροφίας που είναι εφικτή και αηφόρος. Αν έχουμε μεγάλη κλίμακα σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία την εκτατική, μειώνουμε τη δυνατότητα των λιμόνων να συγκρατούν το διοξείδιο του άνθρακος. Είναι αποθετήριο άνθρακος βέβαια οι λιμόνες αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το πώ ακριβώς το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Δεύτερον, ένα μεγάλο μέρος της συζήτηση αφορά τα μεγάλα ζώα, τα βοήδη και τα, σε λιγότερο βαθμό τα εγωπρόβατα. Τι γίνεται όμως με τα, ε, με τα χειροειδή και τα πουλερικά αυτά τρώνε πολλές φορές ε, σόγια ή τρώνε άλλες ε, μορφές ε, τροφίμων δημητριακά κτλ. Εμείς θέλουμε να καλύψουμε λοιπόν όλα τα εκτρεφόμενα ζώα στο σύνολό τους. Εγώ συμφωνώ επίσης με τα πολύ σημαντικά σχόλια που έγιναν από τον αριθμό 34 εδώ μπροστά μας για την ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι όλοι μας έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μια υγιεινή διατροφική δίαιτα. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν πολλές φορές και κορεσμένα λύπη και είναι ανθυγίνα. Είναι απαραίτητο να έχουμε σωστή εκπαίδευση για να επιλέγουμε τα τρόφιμα τα οποία είναι υγιεινά. Κάποιοι άλλοι όμω δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και αυτό είναι άδικο. Θα πρέπει όλοι να έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζήσουν υγιεινά και να διατρέφονται υγιεινά όπως και όλοι μας. Για να απαντήσω τώρα στην ε, εκπρόσωπο της Ένωσης των Γεωργών. Υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την εκτροφή των ε, ζώων και τις εκπομπές από την κτηνοτροφία. Είναι απαραίτητο επίσης να δίνουμε στα ζώα διατροφή η οποία έχει υψηλή ποιότητα γιατί αυτό οδηγεί και σε μεγαλύτερη ποιότητα του κρέατός τους. Και για τους ε, χορτοφάγους οι οποίοι ενοχλήθηκαν ίσως από αυτό το οποίο είπα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ κρέατος και γάλατος, πρέπει να κάνουμε επίσης και μια διάκριση μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών και είναι επίσης πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι φυσικά μπορεί να καλύψει κανείς τις διατροφικές του ανάγκες στις πλούσιες χώρες γιατί υπάρχει δυνατότητα να ενισχύσουμε την διατροφική αξία των προϊόντων. Στις φτωχές χώρες όμως αυτό δεν είναι πάντα δυνατό η πυκνότητα διατροφικών στοιχείων στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι τόσο χαμηλή πολλές φορές που δεν καταφέρνουν οι άνθρωποι να καλύψουν όλες τις διατροφικές τους ανάγκες. Αυτό είναι ένας χώρος έρευνας όπου πλανώνται ακόμα κάποιες αβεβαιότητες αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούν να καλύψουν απόλυτα τις ανάγκες του στις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό θα πρέπει να προωθηθεί όλη αυτή η προβληματική, αυτή είναι η έκκληση που πρέπει να κάνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει το θέμα αυτό σοβαρό, να επανέλθουμε όλοι στις χώρες μας και να θέσουμε επιτάπητο στα θέματα αυτά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι δεν είναι πρόβλημα, θα λυθεί το πρόβλημα των εκπομπών από τι μεταφορέ. θα έχουμε καθαρά αυτοκίνητα κτλ. Όχι, πρέπει να δράσουμε σε όλου του τομεί για να επιτύχουμε του στόχου μα για τα αέρια θερμοκηπίου. Δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό για τον οποίο θα πούν δεν προσπάθησε καθόλου. Yeah, so ευχαριστώ πάρα πολύ για την ζωντανή αυτή συζήτηση και τώρα κάνουμε μια διακοπή για καφέ. Στις 11.30 συνεχίζουμε με το δεύτερο τμήμα της ε, συζήτησης. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ και αυτούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Σε 15 λεπτά τα ξαναλέμε. Μη φέρετε καφέ όμως στην ε, Ολομέλεια σας παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε και πάλι στην συνέχεια της ακρόασής μας για την ε, κλιματική αλλαγή και την διατροφική πολιτική. Λιγότερο κρέας, λιγότερο ζέστη. Ελπίζω να ήταν ε, ευχάριστη διακοπή καφέ και ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε τους υπόλοιπους ομιλητές. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να σας παρουσιάσω τον Ολιβιέ Ντεφούτερ, ο οποίος είναι ο ειδικό εισηγητή για τα δικαιώματα στα τρόφιμα από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών. Πρώτα, όλοι μας προσβλέπουμε σε αυτά τα οποία θα πείτε, για αυτά που πράττει ο Οργανισμός Εθνών για τα θέματα αυτά και για τις συμβουλές που μπορείτε να μας δώσετε. Ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Είμαι ευγνώμων για την πρόσκλησή σας να προσέλθω και να συμβάλλω στην ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις επιπτώσεις των επιλογών μας κατανάλωσης στην ασφάλεια προμήθειας τροφίμων και στο δικαίωμα διατροφής. Γίνεται αυτή η συζήτηση την καλύτερη στιγμή. Πρώτο, διότι είχαμε το 2007 και 2008 την παγκόσμια κρίση των τιμών των τροφίμων και υπάρχει επομένω ένα νέο και άνευ ενδιαφέρον για μια επανεξέταση των, ε, συστημάτων μας παραγωγής ε, τροφίμων, σημαντικές αλλαγές που επίκυνται, οι άμεσες επενδύσεις ε, στην Γεωργία από 3 δις αμερικανικά δολάρια το 2005 έως 2007 φτάσανε μάλλον τότε το 2005 με 2007 στα 3 εκατομμύρια από 600 εκατομμύρια που ήταν στην δεκαετία του 90 είναι μια σημαντική και καλοδεχούμενη εξέλιξη γιατί χρειάζονται τέτοιες επενδύσεις για την μείωση της φτώχειας ένας από τους λόγους για τους οποίους το σύστημα παραγωγής διατροφής περνάει τέτοια κρίση σήμερα είναι διότι από το 1980 οι επενδύσεις στην Γεωργία υπήρξαν πάντοτε ανεπαρκείς όμως δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσα χρήματα πηγαίνουν στην γεωργία, αλλά και για την υποστήριξη ποιων ειδών παραγωγή. Ποιε είναι οι επιπτώσει στα εισοδήματα και ποιε είναι οι επιπτώσει στο περιβάλλον. Δεύτερο, οι κυβερνήσει αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο σήμερα ότι υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ αλλαγών κλίματο και ε, ασφάλειας προμήθειας τροφίμων. Όπω είδαμε πρόσφατα και στην Ανατολική Αφρική, στι Ινδίε, στην Κεντρική Αμερική, στις χώρες εκείνες όπου πλήττονται από το φαινόμενο του Ελνίνιο, η αλλαγή του κλίματος ήδη απειλεί την ικανότητα ολόκληρων περιφερειών, ολόκληρων περιοχών να διατηρήσουν τα σημερινά επίπεδα της αγροτικής παραγωγής. Στην υποσαχαρική Αφρική, αλλά και σε μέρη της Ασίας, η αλλαγή του κλίματος θα επηρεάσει τις βροχοπτώσεις. Θα, αυξηθούν, θα αυξηθεί η περιοδικότητα των ξηρασιών και η μέση ε, ε, θερμοκρασία. Όλα αυτά θα έχουν συνέπειες στην αγροτική παραγωγή. Το, Διεθνέ, το, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή διαπιστώνει ότι μέχρι και 50% θα μειωθούν οι βροχοπτώσεις στην Κεντρική Αφρική από το 2000 μέχρι το 2020 ως αποτέλεσμα της αλλαγής των θερμοκρασιών. Στο σύνολό της η παραγωγική μας ικανότητα σε όλο τον κόσμο θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 3% μέχρι το 2080 σε σχέση με τα επίπεδα του 2000 και μέχρι 16% εάν η θετική επίπτωση του διοξιδίου του άνθρακος στην ε, παραγωγή τελικώς δεν υλοποιηθεί. Και οι, σημαντικές, ε, οι πιο σημαντικές ε, ζημιές θα είναι στην Αφρική και Νότια Αμερική. Είναι αυτά αρκετά σκούρα, αλλά μάλλον αισιόδοξα ακόμη, διότι δεν περιλαμβάνουν τις συνέπειες άλλων γεγονότων όπως πλημμύρες και ξηρασίες, που είναι και οι πιο άμεσες συνέπειες οι εκδηλώσει των αλλαγών του κλίματος. Ούτε λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η αυξανόμε, το αυξανόμενο επίπεδο των θαλάσσιων υδάτων τελικά θα επηρεάσει τους υδροφόρους ορίζοντες τη ξηρά. Επομένως θα μπει αλμυρό νερό στα γλυκά νερά. Λιγότερη επομένως δυνατότητα άρδευση των, γεωργικών, των, των ε, αρρώσιμων γιών. Θα λιώνουν οι μεγάλοι παγετώνε των Ιμαλαίων. Αυτό σημαίνει σημαντικέ. Ε, συνέπειες για την άρδευση και για την υδροδότηση μεγάλων ε, ε, μαζών πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Και επίσης πολλά εκατομμύρια θα, μάλλον ένα δισεκατομμύριο θα πληγεί μέχρι το 2050 και οι σοδιές θα μειωθούν κατά 30% στην κεντρική και νότια Ασία μέχρι το 2050. Επίσης η υποβάθμιση του εδάφους αυξάνεται με τρομακτική ταχύτητα. Είναι θύμα λοιπόν η γεωργία, αλλά είναι και ένοχος. Επομένως, οι άμεσε επενδύσεις στην γεωργία οφείλουν να λάβουν υπόψη και τις συνέπειες ε, στο περιβάλλον. Διότι υπάρχουν συνέπειες οι οποίες αυξάνουν πάλι την ε, ε, αναθέρμανση του κλίματος. η συμβολή της γεωργίας είναι της τάξης 14% στα διοξίδια του άνθρακος. Η χρήση της γης, η αποψήλωση των δασών κλπ. προσθέτουν άλλα 19%. Ναι, μεν τα δάση συγκρατούν το διοξείδιο του άνθρακος και μέχρι 45%, αλλά όπως γνωρίζετε καταστρέφονται σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει ωστόσο ένα ερώτημα το οποίο διαρκώς αποφεύγεται σε διεθνείς συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια προμήθειας τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποιες είναι δηλαδή οι επιπτώσεις των τρόπων κατανάλωσης στις πλούσιες χώρες και ποιες είναι οι συνέπειες στην ικανότητά μας να, τα, να ε, διαθρέψουμε τον πλανήτη. Αυτά είναι σημαντικά ωστόσο και συμβάλλουν στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Τα τρόφιμα που καταναλώνουμε καθορίζουν και με ποιον τρόπο τα παράγουμε. Η αύξηση ε, της ζήτησης προϊόντων ε, κτηνοτροφίας έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται ωστόσο στην τιμή. Από τα 14% των διοξιδίων του άνθρακος που προέρχονται από την Γεωργία, ένα 38% οφείλεται στα λοιπάσματα, 31% στα ε, ζώα που εκτρέφονται και μια μελέτη που λέγεται Livestock Long Shadow, η μακρά σκιά το, της κτηνοτροφίας του 2006, λαμβάνει υπόψη και την αποψήλωση των δασών για να δημιουργηθούν βοσκοτόπια φτάνει σε 18% ε, συμβολή της κτηνοτροφίας ε, στις συνολικές εκπομπές διοξιδίων του άνθρακος, δηλαδή το διπλάσιο των, ε, των μεταφορών. Μαζί λοιπόν βοσκοτόπια, αρρώσιμες γέες, οι γέες που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές φτάνουν στο 70% του συνολικού, της συνολικής γεωρικής γης και 30% όλης της ε, χερσαίας, του χερσαίου πλανήτη. Τα βοσκοτόπια από μόνα τους ευθύνονται για 20-26% και για πολύ περισσότερο στην περιοχή του Αμαζόνιου. Αυτά κυρίε και κύριοι δεν είναι και η καλύτερη χρήση που μπορούμε να κάνουμε των σπάνιων πόρων μας. Το UNEP, το ε, Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, εξέδωσε μια έκθεση για τον ρόλο του περιβάλλοντος στην αποφυγή κρίσεων τροφίμων και λέει ότι μείωση μέχρι το 2050 σε 37,4 κιλά ανακεφαλή της κατανάλωσης ε, προϊόντων ε, κτηνοτροφίας, δηλαδή στο επίπεδο του 2000, θα απελευθερώσει περίπου 400 εκατομμύρια δημητριακών για ανθρώπινη κατανάλωση. Δηλαδή αρκετά για να καλύψουμε τις θερμιδικές ανάγκες 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπων τον χρόνο. Αν συνεχιστούν τα πράγματα όπως είναι, μέχρι το 2050 θα χρειάζονται περίπου 1.573 εκατομμύρια τόνοι δημητριακών για μη, χρήση, για μη τροφική χρήση, από τα οποία τουλάχιστον 1,45 εκατομμύρια τόνοι θα χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές. Αρκετά δηλαδή και να καλυφθούν οι θερμικές ε, ε, ανάγκες περίπου 4,35 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Χωρίς αυτά να είναι τα μοναδικά, οι μοναδικές αρνητικές συνέπειες της ε, εκτινοτροφίας. Η υπερβόσκηση για παράδειγμα και από ζώα όπως αγελάδες, βοηδοί ή ε, έγες. Ε, αφαιρούν από το έδαφος τη δυνατότητά του να ανανεώνεται. Από 720 εκατομμύρια βοηθοί το 1950 έχουμε φτάσει στο 1,5 δις το 2001, σύμφωνα με την ΦΑΟ. Ο αριθμός εγωειδών και προβατοειδών έχουν ε, από, πάει από ένα δισεκατομμύριο περίπου σε ένα δισεκατομμύριο 750 εκατομμύρια στην ίδια περίοδο. Η αύξηση αυτή στην ε, κτηνοτροφική παραγωγή από το 1950 έχει οδηγήσει σε σημαντική υπερβόσκηση παγκοσμίω. Και υπολογίζεται ότι από το 1950 έχουμε χάσει περίπου 680 εκατομμύρια εκτάρια, δηλαδή περίπου 20% των συνολικών παγκόσμιων βοσκοτοπιών λόγω της υπερβόσκησης που τα έχει υποβαθμίσει. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες, γιατί η εικόνα είναι αρκετά περίπλοκη. Τα ζώα που εκτρέφονται στις ε, βιομηχανικές χώρες καταναλώνουν πέντε θερμίδες για κάθε θερμίδα που παράγουν, κρέατος δηλαδή. Στην Ινδία η αναλογία αυτή είναι λιγότερο από μία μισή θερμίδα. Στην Κένια, όπου τα ζώα ε, βόσκουν ελεύθερα, ή εκτρέφονται με παραπροϊόντα της γεωργίας τα οποία δεν μπορούν να καταναλώσουν άνθρωποι, τελικά αποδίδουν περισσότερες θερμίδες από αυτές που καταναλώνουν. Εξάλλου είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η κτηνοτροφία αποτελεί βέβαια και σημαντική πρόσοδο για δισεκατομμύριο περίπου ανθρώπων περίπου ανθρώπων παγκοσμίω και παραπάνω από ένα τρίτο σε γεωργικές περιοχές. Άρα πρέπει να κάνουμε αποδιδουν περισσοτερε θερμιδες απο αυτε των διαφόρων τρόπων παραγωγής κρέατος και σημαντικη προσοδο για ενα δισεκατομμυριο περιπου ανθρωπων παγκοσμιω και παραπανω απο ενα τριτο σε γεωργικες περιοχε αρα πρεπει να κανουμε διακριση αναμεσα των διαφορων τροπων παραγωγη κρεατο και των τρόπων με, τον, με, τον, με τους οποίους αυτές οι παραγωγές επηρεάζουν την ε, παγκόσμια ασφάλεια προμήθειας τροφίμων και με όλες τις αρνητικές συνέπειες όπως ε, τα αρία του θερμοκηπίου, την υπερβόσκηση κτλ. Και αυτά σε διάφορα επίπεδα τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς τρόπους παραγωγής κρέατος και αυτά και στις δύο άκρες του φάσματος και της παραγωγής και της κατανάλωσης. Αυτό που είναι σαφές για μένα είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να καθορίζουμε ποσοτικούς στόχους στην παραγωγή τροφίμων, όπως για παράδειγμα η ανάγκη να αυξηθεί η παραγωγή κρέατος παραπάνω από 200 εκατομμύρια τόνους, ώστε να φτάσει 470 εκατομμύρια τόνους το 2050. Ένα στόχος δηλαδή που έχει οριστεί από τους ε, ε, ειδικού της ΕΦΑΟ την ομάδα υψηλού επίπεδου πριν από την συνεδρίασή τους και ε, το βλέπουν μέχρι το 2050. Και βέβαια με όλα τα προβλήματα για την υγεία που προέρχονται από την αύξηση της κατανάλωσης κρέατος ε, των ανθρώπων. Γι' αυτό και βρίσκω τη σημερινή συζήτηση πάρα πολύ σημαντική. Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να κάνουν πρόοδο μόνο όταν ε, σπάζουν τα ταμπού, όταν οι πιο φωτισμένοι μεταξύ ημών και οι πιο τολμηροί αποφασίζουν να θέσουν ερωτήματα τα οποία άλλοι θα προτιμούσαν να μην ακουστούν ποτέ. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Μπούζεκ και τον αντιπρόεδρο κ. Μακμίλαν Σκοτ για την σύγκληση της παρούσας ακρόασης και αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συνεχίσω τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσους από εσά δεν γνωρίζετε όλο το ιστορικό το μιλητή μας, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο ο ειδικό εισηγητής για τον ΟΗΕ για το δικαίωμα στα τρόφιμα, για τη διατροφή, αλλά ιδρυτής και συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμών για Θεμελιώδη Δικαιώματα και διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου για τη Διδασκαλία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα Πανεπιστήμια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπήρξατε σαφέστατος στα όσα μας είπατε. Πράγματι είναι ανθρώπινο δικαίωμα το δικαίωμα στη διατροφή, το δικαίωμα στα τρόφιμα. Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, ούτω ώστε να έχουν χρόνο να έρθουν να στους ομιλητές άλλοι ομιλητέ και προσβλέπουμε στην συνέχεια. Περιμένετε λίγα λεπτά να αλλάξουμε θέσεις. Uh, Κυρίε και κύριοι, για το τελευταίο τμήμα της ε, ακροάσεώ μας έχουν έρθει δύο υπέρμαχοι της λιγότερη κρεατοφαγία. Και οι δύο είναι χορτοφάγια. Εγώ δεν τρώω κρέας απλώς. Πρώτος ομιλητής μας είναι ο Δόκτωρ Πατσάρη, Όποιος μελετά τα θέματα του περιβάλλοντος και κυρίως το θέμα της αλλαγής του κλίματος γνωρίζει αυτό το θρύλο που είναι πρόεδρος του διακυβερνητικού πάνελ για την αλλαγή του κλίματος, είναι ο Δ. Πατσάρη. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ για την ε, ευκαιρία αυτή. Είναι ένα μεγάλο προνόμιο για μένα να μπορώ να απευθυνθώ σε εσά. Κυρίε και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωση, φίλοι, συνάδελφοι. Είναι πράγματι για μένα μια μοναδική τιμή το να μπορώ να είμαι μαζί σα στην σημερινή αυτή ευκαιρία και να αναφερθώ σε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι κεφαλαίο σημασία για το μέλλον τη ανθρωπότητα και για την ευζοία όλων των ειδών στον πλανήτη μας. Πιστεύω ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής έχει φτάσει πια μια τέτοια έκταση και διάσταση που δεν μπορούμε πια να το παραγνωρίσουμε και να το αγνοήσουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα λάβει χώρα η συνδιάσκεψη της Κοπενχάγης και ελπίζω ότι θα καταλήξει σε μια σημαντική και στεναρή συμφωνία. Όλοι μας λοιπόν μπορούμε να παίξουμε κάποιο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας σε παγκόσμιο επίπεδο σε ένα χρονικό πλαίσιο που να έχει πράγματι κάποιο αντίκτυπο αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς. Πέραν αυτών τα οποία κάνουν οι κυβερνήσεις λοιπόν και οι παγκόσμιοι φορείς, εμείς σαν κοινωνίες, σαν άτομα μπορούμε να πράξουμε πάρα πολλά. Ο Μαχατμα Γκάντι είχε πάντα τη σημαντική αυτή αρχή στη ζωή του, έλεγε να είσαστε ο ίδιος αυτός που ενσαρκώνει την αλλαγή που θέλετε να δείτε και στον κόσμο γύρω σας. Και όταν τον ρωτήσαν ποιο είναι το μήνυμά του για τους άλλους, έλεγε η ίδια μου η ζωή είναι το μήνυμά μου. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε και να μειώσουμε τις επιπτώσεις των προβλημάτων στην κλιματική αλλαγή, αν θέλουμε να μην υπάρξουν αντικές επιπτώσει όχι μόνο στα παιδιά και τα εγγόνια μα αλλά ούτε και στη δική μα ζωή. Πρέπει να κινηθούμε λοιπόν γρήγορα προ την κατεύθυνση αυτή. Θέλω να εστιάσω στο γεγονό ότι η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων είναι ένα τομέα όπου μπορούμε να επιτύχουμε μια σημαντική αλλαγή. Δεν προτείνω κάτι το ριζοσπαστικό, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει όμω να ακολουθήσουμε ένα δρόμο μέσω του οποίου θα μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος από την κτηνοτροφική παραγωγή. Πιστεύω ότι μπορούμε πράγματι να κάνουμε τη διαφορά. Γιατί θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό το, τομέα, γιατί τα 80% των εκπομπών από τη Γεωργία ουσιαστικά προέρχονται από την κτηνοτροφία. Ο ΦΑΟ υπολογίζει ότι περίπου 18% όλων των εκπομπών αερίου και θερμοκηπίου από ανθρωπογενείς δραστηριότητες μέσα σε ένα ορίζοντα 100 ετών προέρχονται από τη δημοτροφία, Γιατί υπάρχουν κάποια αέρια θερμοκηπίου τα οποία έχουν πολύ σύντομη ζωή στην ατμόσφαιρα. Άμα πάρουμε ένα ορίζοντα λοιπόν ενός αιώνα, 9% του διοξιδίου του άνθρακος έρχεται από αυτές τις δραστηριότητες. 37% των αερίων θερμοκηπίου είναι μεθάνιο και 65% είναι οξύδια του αζότου. Υπάρχουν οι εκπομπές λοιπόν και συχνοτροφίας. Υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις. Σύμφωνα με την έκθεση της ΦΑΟ, ο τομέας κτηνοτροφίας είναι ένας από τους δύο πιο σημαντικούς ε, συνεισφορείς στα προβλήματα του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι και η αιστεία της προσοχής μας όταν αντιμετωπίζουμε τα θέματα της υποβάθμισης των εδαφών γιατί και αυτά συμβάλλουν στον κύκλο παραγωγής της κτηνοτροφίας και επίσης σε ό,τι αφορά τη ρήπανση του αέρα και των υδατών. Όλα αυτά επίσης οδηγούν σε μια απώλεια βιοπικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τομέα της κτηνοτροφία, κατά συνέπεια, είναι ο μεγαλύτερο χρήστη εδαφών στον πλανήτη μας. 70% όλων των χρήσεων αγροτικής γης προέρχονται από την κτηνοτροφία και 30% της ε, έκτασης του κόσμου χρησιμοποιείται για κτηνοτροφία. Της ξηράς προφανώς. Υπήρξε στο παρελθόν προσπάθεια πολλών χωρών να αυξήσουν την παραγωγή κρέατος και ζωικών προϊόντων. Για παράδειγμα, 70% της ε, δασικής περιοχής, της πρώην δασικής περιοχής στον Αμαζόνιο καλύπτεται τώρα από λιμόνες και ένα μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κομματιού που έχει αποδασωθεί χρησιμοποιείται για την παραγωγή δημητριακών. Πολλές χώρες στη Λατινική Αμερική στο παρελθόν είχαν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα συναλλαγματικών αποθεμάτων. Αυτό το οποίο φασίσανε είναι να προχωρήσουν σε εντατική παραγωγή ε, βοήου κρέατος εν ώψη της παγκόσμιας ζήτησης και αυτό οδήγησε σε αποψήλωση μεγάλων δασικών εκτάσεων που τώρα έχουν γίνει βοσκότοποι για τα βοηδή και άλλα μεγάλα ζώα. Πρέπει να σας υπενθυμίσω επίσης το θέμα της έντασης της χρήσης ύδατος σε αυτές τις δραστηριότητες. Ένα κιλό κρέατος χρειάζεται περίπου 1.300 λίτρα νερό, 900 λίτρα για τα, ε, για τα πουλερικά, 4.800 για τα χειροειδή και για τα βοηδή 1500 λίτρα. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε τεράστια πίεση στους υδάτινους πόρους πολλών περιοχών του κόσμου. Το Διεθνές Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή προβλέπει ότι στην Αφρική μέχρι το 2020 θα έχουμε από 75 έως 250 εκατομμύρια άτομα που θα έχουν πρόβλημα να έχουν υδάτινους σπόρους λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε την αντιδικοποίηση της ε, παραγωγής κρέατος και αυτό φυσικά επιδεινώνει τα προβλήματα της πίεσης για την εξέβρεση υδατινών πόρων. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός ανθρώπων στον πλανήτη μας που υποσυτίζονται, που δεν έχουν αρκετή επαρκή διατροφή ενώ παράλληλα ένα μεγάλο μέρος των δημητριακών που παράγονται σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές. Εάν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ε, δημητριακών θα βοηθούσε την παγκόσμια τροφιμική ασφάλεια και θα εξασφάλιζε καλύτερη διατροφή σε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων στο πλανήτη μας. Ένα τρίτο τα εκατό των ε, δημητριακών σε παγκόσμιο επίπεδο και πάνω από 90% της σόγιας που παράγεται χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές. Αυτά είναι τεράστια, τεράστιες ποσότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων και όχι των ανθρώπων. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εγγενής έλλειψη αποτελεσματικότητας στην παραγωγή κρέατος. Χρειάζονται πάνω από 10 κιλά ε, ζωοτροφών, ουσιαστικά δημητριακά, για να παραγάγει κανείς ένα κιλό κρέατος. Αυτή είναι η έλλειψη αποδοτικότητας. Αν το αν τα συγκρίνετε με την σόγια, η, τα στέικς από τόφου είναι 10 φορές λιγότερο εντατικά στην εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος σε ό,τι αφορά την παραγωγή τους. Επομένως, η λιγότερη κατανάλωση κρέατος, το τονίζω αυτό σε ακροατήρια σε όλο τον κόσμο, τονίζω ότι το να μειώσει κανείς την, την, την κατανάλωση κρέατος είναι καλό όχι μόνο για το περιβάλλον και τον πλανήτη μας, αλλά και για την ανθρώπινη υγεία. Χαίρομαι ιδιαίτερα ότι στην χώρα που βρίσκομαι εδώ, πριν από ένα μήνα ήμουνα στη Γάνδη και έδωσα μια ομιλία και από αυτή την ομιλία ξεκίνησε μια κίνηση ώστε μία μέρα τη βδομάδα να είναι μια μέρα χωρίς κρέας. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να υποστηρίξω είναι αυτό το οποίο έχει τονίσει ο Πολ Μακάρτνη εδώ και πολύ καιρό ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε μια μέρα κάθε εβδομάδα και να είναι μια μέρα που να μην καταναλώνουμε καθόλου κρέας. Σήμερα υπάρχουν 20 δισεκατομμύρια ζώα σε αγροκτήματα και πουλερικά τα οποία εκτρέφονται. 250 τόνοι κρέατος παρήχθησαν το 2006, πέντε φορές περισσότερο από τις δεκαετία του 1950. Και παρόλα αυτά οι πατέρες μας και οι παππούδες μας ήταν εύρωστα άτομα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο θα πρέπει να θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η ζωική πρωτεΐνη για να εξασφαλίσουμε άτομα τα οποία θα είναι υγιή. Και εξάλλου, όταν αντιμετωπίζω τέτοιους ισχυρισμού, τους λέω ότι υπάρχουν δύο ειδικοί που θέλω να τους, ε, οποίους θέλω να σας ε, παραπέμψω που είναι ειδικοί σε χορτοφαγικές ε, δίαιτες. Είναι τα άλογα και οι ελέφαντες που όλη τους η διατροφή βασίζεται σε φυτικά προϊόντα. Και θέλω να κλείσω την παρέμβασή μου λέγοντας ότι ένας μεγάλος αριθμός ε, διακεκριμένων ατόμων έχουν ακολουθήσει χορτοφαγικές δίαιτες. Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν είπε ότι τίποτα δεν θα βοηθήσει περισσότερο την ανθρώπινη υγεία και την διατήρηση της ζωής στον κόσμο όσο η πορεία προς μια χορτοφαγική δίαιτα. Και αυτό τώρα έχει αποδειχθεί από έρευνα η οποία έχει δημοσιευθεί στο Lancet, το ιατρικό περιοδικό, και θα ακούσατε και περισσότερο για αυτά τα θέματα. Ο Λέων Τολστό είπε ότι αν κάποιο θέλει να ζει με δίκαιο τρόπο, πρέπει καταρχήν η πρώτη του αποχή να είναι από τα ζωικά προϊόντα και ο Σερ Πολ Μακάρνι, ο οποίο θα πει πολύ περισσότερα, τον παραθέτω, είπε ότι η χορτοφαγία αντιμετωπίζει πάρα πολλά πράγματα μαζί, την οικολογία, τα, θέματα, τα προβλήματα του λοιμού και την βία προς τα ζώα. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι κυρίως από την έποψη της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής αυτός είναι ένας απλός και αποτελεσματικός κανόνας, ένα απλό μέτρο που όλοι μας μπορούμε να υποστηρίξουμε και να εφαρμόσουμε με το δικό μας τρόπο. Δηλαδή για να βοηθήσουμε τις μελλοντικές γενιές να μην υποστούν τις αντικές συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Εν κατακλείδη, αν συνεχίσουμε στο δρόμο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, το σενάριο business as usual, τότε ο αντίκτυπος κλιματικής αλλαγής, όπως είπα και στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου, παρόν των 100 περίπου και παραπάνω αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, όλα αυτά θα οδηγήσουν σε τρομερή διαταραχή της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής σε πάρα πολλά τμήματα του κόσμου. Η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι υπάρχει ένας κίνδυνος πάνω από 10 ή 12 κράτη να γίνουν αποτυχημένα κράτη μέσα σε εισαγωγικά, κάτι το οποίο θα έχει επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής και στις κοινωνίες μας. Γιατί αυτές είναι οι κοινωνίες οι οποίες προωθούν το λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών, την τρομοκρατία και την παράνομη μετανάστευση. Τα κράτη αυτά τα αποτυχημένα, επομένως όλοι έχουμε ένα καθήκον να δράσουμε για να προστατεύσουμε το κλίμα του πλανήτη μας και να μειώσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας σε 2 βαθμούς Κελσίου το πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να περιορίσουμε την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και σας τονίζω και πάλι ότι η μείωση της κατανάλωσης κρέατος θα είναι ένας πάρα πολύ αποτελεσματικός στόχο, τρόπος να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτά που είπατε και για όσα κάνετε. Είπα ότι ο μιλητής μας ήταν ένας θρύλος Ο Σερ Πολ Μακάρτνε είναι κάτι παραπάνω από θρύλος Είναι ένα υπέρλαμπο αστέρι. Και διακόπτει το, την τουρνέ του στην Ευρώπη. Έπαιζε χθε το βράδυ στο Αμβούργο και επιστρέφει στο Βερολίνο απόψε. Και διακόπτει για να έρθει εδώ. Τον ευχαριστώ όχι μόνο επειδή ήρθε, αλλά διότι δίνει και χρόνο και ενέργεια για ένα θέμα στο οποίο πιστεύει και εκείνος και εγώ. Δηλαδή ότι όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε ο καθένας ξεχωριστά στη μείωση της άξιας τρώγοντα τρώγοντας λιγότερο κρέας. Ο Πολ έγραψε το πιο δημοφιλές τραγούδι στον κόσμο, το Yesterday. Σήμερα μιλάει για το αύριο. Έγραψε το τραγούδι για το χθε, σήμερα μιλάει για το αύριο. Το αύριο το δικό σα και των παιδιών σα. Σερ Πολ Μακάρτιν, έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε εδώ σήμερα. Μιλώ εκ μέρου τη εκστρατεία που ξεκινήσαμε στον Ηνωμένο Βασίλειο. Μια Δευτέρα χωρί κρέα είναι ο τίτλο τη εκστρατεία. Πώ εκλήθη να συμμετάσχω σε αυτή την εκστρατεία. Διάβασα μια ιστορία για την έκθεση του ΟΗΕ. Έκθεση που εκδόθηκε το 2006 που ε, ήταν η μακρά σκιά της κτηνοτροφίας ήταν ο τίτλος δεν το έγραψε, δεν έγραψε την έκθεση κάποιο χορτοφάγο. Αν είχαν γράψει την έκθεση οι χορτοφάγοι, ε, θα λέγανε φυσικό είναι το οποίο αυτό ένα χορτοφάγο. Αλλά εκείνοι που έγραψαν την έκθεση στο ΟΗΕ, πιθανότατα ήταν ε, άνθρωποι κανονικοί, που έτρωγαν παραδοσιακά ε, τρόφιμα και έτρωγαν κρέα οι ίδιοι. Αυτό με προσήλκησε. Άρχισα να στέλνω κάποια γράμματα στου αρχηγού κρατών και του έλεγα αυτό θα θεωρείτε ότι εγώ είμαι ένα κορτοφάγο που χτυπάω την πόρτα σα για να μιλήσω για το επιμένο μου θέμα. Αλλά του είπα ότι αυτό που βλέπετε το έγραψα εγώ. Και αυτά είναι στοιχεία που συνέλεξε ο ΙΕ. Έκτοτε, πολλές μελέτες και εκθέσεις έχουν εκδοθεί στο New York Times και στους Times του Λονδίνου πρόσφατα, στα πρωτοσέλιδα, με το θέμα αυτό Πιστεύω προσωπικά ότι υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη. Όπως είπε και ο Δόκτωρ Μπατσάρη, η βιομηχανία εκτινοτροφική παράγει περισσότερα έργα θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών, από τις μεταφορές μαζί. Τρένα, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, φορτηγά. Και εμείς θεωρούμαστε ότι ήμασταν οι κακοί αλλά φαίνεται τελικά ότι η κτηνοτροφία παράγει περισσότερα αέρια θερμοκηπίου. Μιλάμε και για τον αποψήλωση των δασών. Έξι γήπεδα ποδοσφαιρικά εξαφανίζονται κάθε λεπτό δασών, στην αποψήλωση των δασών, για να βοσκούν τα ζώα ή να παράγονται ε, κτηνοτροφές. Νερό για ένα μπέργκερ χρειάζεται εξίσου τόσο νερό όσο χρειαζόμαστε για να κάνουμε ένα ντους για τέσσερις ώρες. Αυτά είναι ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα χαιρόμουν αν όλα αυτά δεν ήταν αληθή, διότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε επάπειρον όπως ζούμε τώρα, να είμαστε ικανοποιημένοι και να μην ασχολούμαστε με το θέμα. Αλλά αρχίζω να αισθάνομαι ότι αληθεύουν όλα αυτά και είναι άσχημο συνέστημα και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. 8% της χρήσεως νερού στον κόσμο οφείλεται στην κτηνοτροφία. Και η κτηνοτροφία είναι μεγαλύτερη πηγή ρήπανσης των υδάτων. Ορμόνες, αντιβιωτικά, χημικά, από εκεί πηγαίνει γίνεται εξαρτησία των δεμάνων και λοιπά, παρασιτοκτόνα, λιπάσματα, τα απόβλητα των ζώων. Οι ζωοτροφές επίσης αφήνουν πάρα πολύ μεγάλο ίχνος άνθρακα όσον αφορά τη μεταφορά τους και τη χρήση γεών. Ένα τρίτο από τα δημητριακά που καλλιεργούνται, καλλιεργούνται για να τρέφουν τα ζώα και 90% της όγια που καλλιεργείται είναι για να τρέφει τα ζώα χρειάζεται 40 θερμίδες ορυκτών καυσίμων για να παραχθεί μια θερμίδα ε, ενός ε, βοηού κρέατος. 2,2 θερμίδες για να παραχθεί μια θερμίδα μιας πρωτεΐνης φυτικής. Πάμε τώρα στις εκπομπές από τα ζώα, από της κτηνοτροφίας. Επειδή δουλεύει έτσι στο μάχη της Αγελάδας, ξέρουμε ότι είναι μυρικαστικό. Άρα αναγκάζονται να ρευτούν Οπότε παράγουν μεθάνιο. Θα ξέρετε αυτά τα γεγονότα, αλλά πρέπει να τα επαναλάβουμε. Το μεθάνιο, κάθε μόριο μεθανίου, έχει 21 φορές περισσότερη δύναμη παγίδευσης θερμότητας από ότι το διοξείδιο του άνθρακος και μένει στην ατμόσφαιρα 9 με 15 χρόνια. Πολύ μεθάνιο μένει. Αυτό ήταν στο Science World του 2002. Η κτηνοτροφία παράγει και πολλά οξύδια του αζότου. 310 φορές πιο ισχυρό είναι αυτό και παραμένει στην ατμόσφαιρα 114 χρόνια. Τα αέρια λοιπόν που απελευθερώνται σήμερα θα επιδεινώνουν το κλίμα επί σειρά δεκαετιών στο μέλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος για το τι μπορεί να κάνει. Ο κόσμος θέλει να κάνει κάτι, θέλει να κάνει τη διαφορά, δεν ξέρει όμως πώς, τι να κάνει, τι λέει εξατία μας. Προσπαθήστε να έχετε μία μέρα την εβδομάδα που έντοτε κρέας. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Και είναι ενδιαφέρον αν το ψάξει κανείς. Προτείνουμε μία Δευτέρα χωρίς κρέας, βέβαια μπορεί να διαλέξετε μία οποιαδήποτε άλλη μέρα. Περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτό που με τραβάει σε αυτή την ιδέα είναι ότι είναι εφικτό, εύκολο να το κάνει. Αν πει στον κόσμο, γίνε χορτοφάγο, αυτό είναι πολύ δύσκολο για του περισσότερου να γίνουν χορτοφάγοι. Χρειάζεται να έχει πάθο. Να, να προβληματίζεται, να θέλει να το κάνει. Αλλά αν πει στον κόσμο, μία μέρα. Οι περισσότεροι κάπου το έχουν ρίξει έξω το Σαββατοκυριακό και τη Δευτέρα θα να πάνε στο γυμναστήριο. Οπότε θα μπορούσαν να μην φάνε κρέα εκείνη την ημέρα. Ίσως να είναι μια καλή μέρα να διαλέξουν να το κάνουν αυτό. Ε, παλιά δεν ανακυκλώναμε, δεν μας ενδιαφέρει η ανακύκλωση, αλλά τώρα έχει γίνει αποδεκτή ανακύκλωση. Στην καθημερινή μας ζωή, στα υβριδικά αυτοκίνητα δεν τραβούσαν τον κόσμο. Αλλά σήμερα είναι πολύ δημοφιλή. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δώσουμε μια απάντηση στον κόσμο. Λοιπόν, προτείνω, μία μέρα της εβδομάδας χωρίς κρέας θα περικόψει τις εκπομπές και θα μειωθεί αντίστοιχα με το όσο θα κατανάλωνε ένα, θα εξέπεπε αυτοκίνητο για να κάνει ένα ταξίδι χιλίων μιλίων. Τόσο θα ήταν η μείωση. Έχουμε το παράδειγμα της Γάνδης που έχει μια μέρα χωρίς κρέας. Στις ΗΠΑ η Βαλτιμόρη. Έχει σχολικό σύστημα όπου εκεί 80.000 παιδιά δεν τρώνε κρέας μια μέρα την εβδομάδα. Σουηδία. Άρχισαν να βάζουν ετικέτες στα τρόφιμα και να δείχνουν στους καταναλωτές ποια είναι η περιβαλλοντική συνέπεια που προξενεί αυτό το τρόφιμο. Διαλέγει ο άνθρωπος δηλαδή. Σου λένε ότι αυτό το μπέργκερ, αυτό το μπιφτέκι θα βλάψει την ατμόσφαιρα κατά τόσο. Οπότε ο πελάτης μπορεί να δει το προϊόν και να πει ίσως δεν θέλω να το αγοράσω αυτό. Οπότε ο καταναλωτής μπορεί να αγοράζει υπεύθυνα και λογικά. Στο Σάο Πάολο, στην Βραζιλία, διότι η Βραζιλία είναι τεράστιος εξαγωγιάς κρέατος και εκεί έχουν μια μέρα που δεν τρώνε κρέα. Και στον Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν αρκετά σχολεία όπου εκεί ακολουθούν αυτή την εκστρατεία. Και μία ε, διευθύντρια μου είπε ότι ανησυχούσε ότι οι γονεί ίσω να θεωρούσε ότι έδινε πολιτική χρειά στο θέμα, όπω το παρουσίασε τα παιδιά. Αλλά τελικά δεν ανησύχησαν οι γονεί μου, είπε η γυμνασιάρχησα, διότι όλοι θέλουν να κάνουν κάτι και αρέσει πολύ στα παιδιά, διότι είναι το μέλλον του. Θεωρούμε ότι επειδή τα παιδιά είναι μικρά, ότι είναι ανόητα. Δεν είναι όμω. Δεν είναι κουτά. Καταλαβαίνουν ότι είναι ο πλανήτη του. Θα κληρονομήσουν αυτόν τον πλανήτη. Και αν τον αφήσουμε στα χάλια του, θα πρέπει να καθαρίσουν την όλη κατάσταση. Οπότε συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα παιδιά καταλαβαίνουν το πρόγραμμα, ενστερνίζονται την ιδέα, είναι ο πλανήτης τους αυτού. Και σαν γονείς όλοι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά μας. Πικιλοτρόπος. Έτσι πρέπει να δούμε τι ευθύνε έχουμε έναντι του μέλλοντο. Πρέπει να υπομιστούμε τι ευθύνε του μέλλοντο των παιδιών μα. Και όπως είπε και ο δόκτωρ Πατσάρη, η υγεία είναι η άλλη πτυχή του θέματος το, ο ερευνητικό φορέα το καρκίνο ε, στον κόσμο είπε ότι πρέπει να καταναλώνουμε λιγότερο ερυθρό κρέα. Και αυτό αφορά λοιπόν την υγεία και των παιδιών και των ενηλίκων. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσει του, του κόσμου. Εγώ προτείνω ότι ίσω θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν και να κατευθύνουν τον κόσμο να μειώσει την κατανάλωση του κρέατο. Διότι τώρα νέα ηθικά θέματα έχουν ανακύψει. Και δεν είναι πολύ ηθικό να αγνοεί αυτά τα ζητήματα δεν είναι πλέον προσωπική επιλογή αυτή που συζητάμε. Είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει όλο τον πλανήτη. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε έτσι. Όμως όταν προκύπτει μια κρίση ή προέκυψε κάτω παρελθόν, τα κοινοβούλια και οι λαοί αντιμετώπισαν το θέμα. Άρα μπορεί κάτι να γίνει. Παραδείγματο χάρη, σκεφτείτε το εξή. Στο Λονδίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια ή στο Λο Άντζελε. Στο Λονδίνο από ό,τι ξέρω. Όταν μεγάλωνα εφημερίδε κάθε χειμώνα είχα μια φωτογραφία της εθαλομίχλης του Λονδίνου, το smog, την ομίχλη ε, και λέγανε ότι ήταν ο ατμός της, σαν ένα ατμός της σούπας που μαγείρε ε, ε, και δεν μπορούσε να δει τίποτα και λέγανε ότι είναι κάτι απλό αλλά εμείς δεν βλέπαμε αλλά όταν είδαν ότι αυξανόταν η θανάτη, η θάνατη και διαπίστωσαν ότι κινδύνευε η υγεία και καθαρίσαν το Λονδίνο. Σήμερα είναι καθαρό το Λονδίνο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Έπρεπε να γίνει κάτι, έγινε κάτι. Ε, το κάπνισμα στο δημόσιο χώρο. Εγώ μεγάλωσα σε ένα δωμάτιο γεμάτο καπνό. Σε κάθε οικογενειακό πάρτι όλοι κάπνιζαν. Και εγώ δεν θεωρούσα ότι κάτι έτρεχε. Και οι δύο γονεί μου, ε, και οι δύο κάπνιζαν, η, ε, η μητέρα μου πέθανε από καρκίνο. Εγώ δεν θεωρούσα ότι ήταν πρόβλημα το κάπνισμα και εγώ επί μεγάλο χρονικό διάστημα κάπνιζα. Αλλά από τη στιγμή που οι γιατροί είδαν ότι το κάψιμο συνδέεται με πολλές ασθένειες και γνωστοποιήθηκε και το παθητικό κάπνισμα, έπρεπε κάτι να κάνουμε, πρέπει να κάνουν κάτι οι κυβερνήσει. Και τώρα δεχόμαστε ότι κανένα δεν μπορεί εδώ σε αυτή την αίθουσα να καπνίσει, πρέπει να βγει έξω. Το δεχτήκαμε αυτό. Ήταν τεράστια αλλαγή, δεν ήταν δημοφιλή, αλλά έπρεπε κάτι να γίνει. Για το μέλλον του πλανήτη λοιπόν οι κυβερνήσεις και το κοινοβούλιο σε αυτή την περίπτωση μπορούν να ενθαρρύνουν και να ενημερώσουν και να βοηθήσουν τον κόσμο να δει πόσο εύκολο θα ήταν κάποιος να μην φάει κρέας για μια μέρα. Και κάτι άλλο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Να βοηθήσουμε και τους αγρότες. Διότι αυτό είναι κάτι που συνέχεια βλέπουμε μπροστά μας. Αν έχουμε λιγότερα ζώα στην κτηνοτροφία θα πληγούν οι ε, κτηνοτρόφοι. Αλλά οι κυβερνήσει και τα κοινοβούλια πρέπει να βοηθήσουν του γεωργού, του κτηνοτρόφου να ακολουθήσουν νέε πρακτικέ, να προσαρμοστούν. Αυτό έγινε καθ' όλη τη διάρκεια τη ιστορία. Έπρεπε να γίνουν αλλαγέ. Έπρεπε να αλλάξουν τον τρόπο τον οποίο κάναμε τα πράγματα. Και νομίζω ότι τώρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη να κάνουμε και άλλη αλλαγή. Πρέπει να εξηγήσετε στου γεωργού τι μπορούν να καλλιεργούν, πώς μπορούν να πετύχουν τα ίδια επίπεδα παραγωγικότητας, αλλά με διαφορετικό τρόπο θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Εγώ ο ίδιος ζω σε μια εκμετάλλευση βιολογικής παραγωγής και όταν δέκα χρόνια αποφασίσαμε τη βιολογική παραγωγή όλοι γύρω μου λέγανε τι είναι αυτός, χαζός είναι. Ε, δεν έχει νόημα, δεν θα πετύχει και τώρα δεν το λένε αυτό συμφώνησαν, ε, το, το έχουν εστερνιστεί, είναι καλές οι τιμές για τα βιολογικά προϊόντα και πολλοί από αυτούς αλλάζουν και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό. Εδώ τι σας προτείνω σήμερα, γι' αυτό είμαι εδώ. Να σας πω ότι το πρώτο βήμα είναι μια μέρα της εβδομάδας χωρίς κρέας, μια Δευτέρα χωρίς κρέας. Να συνηθίσουν οι άνθρωποι την ιδέα. Δεν είναι νέα ιδέα. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί και κατά το παρελθόν. Ο πρόεδρος Τρούμαν το 1947 στην πρώτη τηλεοπτική του ομιλία προς τον Αμερικανικό λαό μίλησε για την κρίση στην Ευρώπη και προς ο Αμερικανικός λαός θα πρέπει να βοηθήσει μετά τον πόλεμο ήταν αυτό και ότι έπρεπε να δώσουν βοήθεια υπό τη μορφή τροφίμων και τι πρότεινε το 1947 πρότεινε να μην φάνε κρέας την Τρίτη και προχώρησε πιο πέρα και πρότεινε την Πέμπτη να μην φάνε πουλερικά και αυγά και αυτό ήταν κάτι που συνέβη. Το ξεχνάμε αυτό. Αυτό έγινε. Έχει σημειωθεί στην ιστορία. Πρέπει να δούμε και την φτώχεια στον κόσμο. Όπου εκεί έχουμε 1,4 δις ανθρώπους που ζουν σε μεγάλη φτώχεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα. Και ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε την κατανάλωση του κρέατος. Μύρισα στον Αλ για αυτό το θέμα. Είναι πολύ γνωστός ο Αλγκόρ για τις απόψεις που έχει όσον αφορά την αύξηση θερμοκρασίας. Και τον ρώτησα και του λέω θα μπορούσε να μου δώσει μια δήλωση να σας διαβάσω σήμερα. Και είχε την καλοσύνη να μου δώσει μια δήλωση. Λέει, ανάμεσα στα αίτια της κρίσης της κλιματολογικής είναι η μεγαλύτερη ε, κατανάλωση κρέατος στον κόσμο. Κυρίως όταν τα ζώα μεγαλώνουν με επιζήμιους τρόπους της εκμεταλλεύσεις. Παίρνουν από τους, από τους τα ζώα. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η λιλεπίδραση μεταξύ ζώων και φυτών. 6.000 γαλόνια για κάθε λίβρα πρωτεΐνης χρειάζεται. Και παράγονται πολλά απόβλητα ε, όξινα από τα ζώα και θα πρέπει τα απόβλητα των ζώων αντί να επεξεργάζονται ε, κανονικά, επεξεργάζονται σαν τοξικά απόβλητα και δημιουργούν προβλήματα στην περιοχή που βρίσκονται. Εγώ δεν είμαι χορτοφάγο, λέει ο Αλγκόρ, αλλά δέχομαι τι ιατρικέ ενδείξει ότι η αύξηση κατανάλωση ερυθρού κρέατο στον κόσμο συνδέεται επίση με την αυξανόμενα ποσοστά ασθενειών, ε, καρδιακών ασθενειών, καρδιακιακών ασθενειών. Για όλου αυτού του λόγου, οι πρωτοβουλίε που έχουν στόχο να μειωθεί αυτή η τάση, όπω να μην τρώει κανεί κρέα την Δευτέρα, είναι υπεύθυνε ευπρόσδεκτε συνιστώσει μια γενική συνολική στρατηγική για την μείωση τη ρήπανση και μείωση τη αύξηση θερμοκρασία και βελτίωση ταυτόχρονα τη ανθρώπινη υγεία. Λοιπόν, συνοψίζοντα, σα παροτρύνω τον καθένα από εσά να κάνετε αυτό που μπορείτε για τους λαούς σας, για τα παιδιά του και για τον πλανήτη που θα κληρονομήσουν. Λοιπόν, να έχουμε μία μέρα χωρίς κρέας, μία Δευτέρα χωρίς κρέας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πολ. Είτε συμφωνείτε, είτε διαφωνείτε. η πρόθεσή μου σήμερα ήταν να εστιάσουμε την προσοχή σας στο θέμα της κτηνοτροφικής παραγωγής, της κατανάλωσης κρέατος, του αντίκτυπού του για την ανθρώπινη υγεία και φυσικά και για το περιβάλλον. Ο Σερ Πολ, όπως και πολλοί άλλοι, έχουν υπογράψει μια κοινή δήλωση για να κλείσουμε αυτή τη συνεδρία και να σας διαβάσω. Είμαστε ευγνώμονες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτήν την ε, συνδιάσκεψη, για την ακρόαση με την ευκαιρία και τη ε, συνθήκη Λισαβόνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει πιο μεγάλη ευθύνη μαζί με τι κυβερνήσει να προωθήσει πρωτοβουλίε σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπίσει προβλήματα του περιβάλλοντος και ιδίω να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Ζητούμε λοιπόν από τους βουλευτές να βοηθήσουν σε αυτό τον αγώνα με το να καταναλώσουν και ε, λιγότερο κρέας. Πρόκειται για τον Σερ Πολ Μακάρτη, τον κύριο Πατσάουρη και εμένα. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να αναπτύξουμε πολιτικές περιβάλλοντος, πολιτικές ε, δημόσιας υγείας που να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της κτηνοτροφίας σε επίπεδο, σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής. Ζητούμε από τις κυβερνήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες και τους Δήμους να κάνουν αυτή την έκκληση για τη μείωση κατανάλωσης κρέατος από τους ε, εργαζόμενους, αλλά ζητούμε και από όλους να αλλάξουν τη δίαιτά τους και να έχουν μία ημέρα χωρίς κρέας την εβδομάδα, ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος. Συνάδελφοι, φίλοι, έχουμε κάνει ειδικέ ρυθμίσεις σήμερα στα, στις καφετέρες και τα εστιατόρια του Κοινοβουλίου τα μισά πιάτα τα οποία διαθέσιμα θα είναι χωρίς κρέας. Και αυτό είναι μια πρώτη εκκίνηση αν θέλετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς λοιπόν που είναι παρόντες εδώ, τους ομιλητές, όλο το προσωπικό που συνέβαλε σε αυτήν την ε, συνεδρίαση, αλλά ιδίως στους δύο τελευταίους ομιλητές, τον κύριο Ρατζέντα Πατσάουρη και τον Σερ Πολ Μακάρντ. Ευχαριστώ.